die Präsidentin. Herr Giegold ist jetzt ganz erschrocken. Τρόμαξε ο κύριος Γκίγκολτ από τη Φέντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι που είστε παρόντες, ε, άρχεται η συνεδρίαση. Και θα ξεκινήσουμε πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έκθεση της κυρίας Ιντφέλντα το πανευρωπαϊκό ε, προϊόν συνταξιοδότησης. Κυρία Ιντφέλντ, ως εισηγήτρια, έχετε το λόγο τα λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ε, κύριε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι που σήμερα θα μπορέσουμε επιτέλους να ψηφίσουμε το ΠΕΠ, όπως το αποκαλούμε, το Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν διότι νομίζω ότι τα καταφέραμε να σας παρουσιάσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό προϊόν που θα είναι απλό και ασφαλές για τους καταναλωτές. Αυτό νομίζω ότι έχετε μπροστά σας. Πρώτα απ' όλα είναι πανευρωπαϊκό. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος καθορίζει πανευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας και δικαιώματα για τους καταναλωτές, αλλά επίσης και πανευρωπαϊκή επιτήρηση του προϊόντος, τη δυνατότητα του ΕΙΟΠΑ να παρέμβει. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αρχικά θέλαμε να υπάρξει έγκριση του προϊόντος από το ΕΙΟΠΑ, αλλά με την ευφύ χρήση των υφισταμένων αρμοδιοτήτων του ΕΙΟΠΑ επιτύχαμε τον ίδιο στόχο. Επίσης καθορίσαμε αναλυτικά τα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών, το δικαίωμα να λάβουν ενημέρωση, υποχρεωτική συμβουλή, το δικαίωμα να αλλάζουν προϊόντα, την φορητότητα του προϊόντος. Επίσης επιτύχαμε το ανώτατο όριο του κόστους να είναι 1% και αυτό δεν ήταν εύκολο γιατί υπήρξε τρομερά έντονη αντίδραση και αν δείτε τώρα ποιο είναι το κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων το ανώτατο όριο 1% είναι πολύ καλό επιτύχαμε ένα προϊόν βάσης που θα είναι έτοιμο παράδοτο και για άτομα που δεν γνωρίζουν πολλά για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και που δεν είναι ιδιαίτερα ε, ευκατάστατα, ούτως ώστε να έχουν ένα χρήσιμο προϊόν. Είδαμε πρόσφατα όμως ότι πολλοί ακόμη έχουν ανησυχίες και θα ήθελα να ε, αντιμετωπίσω μας παρανοήσεις. Το ΠΕΠ e είναι προϊόν τρίτου πυλώνα σαφώς. Είναι συμπληρωματικό, ατομικό και εθελούσιο. Δεν αντικαθιστά τα προϊόντα πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Γιατί πήρα πολλά email, όπως και περισσότεροι συνάδελφοι υποθέτω, ιδιαίτερα από την Ισπανία, που μας κατηγορούν ότι καταστρέφουμε το δημόσιο συνταξιδοτικό σύστημα. Αλλά αυτά είναι ανοησίες. Και θέλω να πω ότι ο μόνος πραγματικός κίνδυνος προς ε, το δημόσιο συνταξιοδοτικό είναι οι εθνικές αρχές που είναι ε, που δεν είναι σε θέση και δεν επιθυμούν να μεταρρυθμίσουν τα συστήματά του Το ΠΕΠ θα συμπληρώσει τις ε, συντάξεις εκεί που είναι ανεπαρκής και που είναι ανεπαρκής φταίνει οι εθνικές κυβερνήσεις και όχι το ΠΕΠ. Θα δώσει τη δυνατότητα σε όσου εργαζόμενους δεν έχουν σωστή συνταξιοδοτική κάλυψη σήμερα να έχουν κάτι για τα γερατιά τους. Επίσης, η δημιουργία ενός τέτοιου προϊόντος ε, καλού για τους καναλωτές ήταν ε, η πρωταρχική μου ανησυχία, το πρωταρχικό μου μέλημα. Και ξέρω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συμπληρώσει, να ολοκληρώσει την ε, κεφάλαια αγορά. Δημιουργούμε κάτι που είναι καλό για τους πολίτες μας, που ήταν ο βασικός μας στόχος. Οπότε αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε σήμερα θα επιτύχει αυτό το στόχο και θα συμβάλλει περαιτέρω στην οικοδόμηση της κοινωνικής Ευρώπης που φροντίζει τους πολίτες της και ελπίζω να εγκριθεί με ευρία πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Ο κύριος Κατάινεν, παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, οργάνωση αυτής της ε, συζήτησης για το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Στεξιωτικό Προϊόν. Πρόκειται εδώ για μια πρόταση που αποτελεί ορόσημο στην κάλυψη των ε, κενών στα στεξιωτικά συστήματα και τη δημογραφική εξέλιξη. Ένα προϊόν το οποίο θα είναι ωφέλιμο για το καταναλωτή. Μια πρόταση η οποία θα εξασφαλίσει ένα πλαίσιο με ισχυρή προστασία του καταναλωτή και με ενίσχυση της του διασυνοριακού ανταγωνισμού. Όπως είπε και η συγκήτρια, δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα συστήματα ταξιοδότησης. απλώς συμπληρώνει εκείνους που θα ήθελαν να έγραφουν στο σχέδιο αυτό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νιτφέλτ, την εισηγήτρια, η οποία αφιέρωσε πολύ χρόνο αλλά και με πολύ πάθος ε, συνέβαλε στην υλοποίηση του ΠΕΠ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Γκουαλτιέρη, πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ, τους, τους κύριους Χέις, Σόρο, Άικχουτ, Κόξ, Άνεμενς, Ντίκουμ, σκιώδεις ηγητές για την επικοδομητική του συνεισφορά για την επιμονή και για την πίστη που έδειξαν σε αυτή την ε, μεγάλη πρόκληση. Και επίσης όλους τους ε, συνεισηγητές από την ε, ΕΚΟΝ και την ΕΜΚΟ που συνέβαλαν τα μάλλα. Οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που από τώρα μέχρι το 2057 θα ε, θα, θα δουν μια εξοικονόμηση σημαντική και βεβαίως ε, με δεδομένο τον κατακαιρματισμό της αγοράς των συνταξιδοτικών ταμείων, ανυπαρξία μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί 67 μόνο από τα 243 εκατομμύρια των πολιτών μεταξύ των 25 και 59 ετών ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει επενδύσεις σε ένα συνταξιωτικό σύστημα. Έτσι λοιπόν με το νέο αυτό σύστημα θα μπορούν σε καθαρά εθελοντική βάση να οργανώνουν τη σύνταξή τους με ένα μοντέλο που θα συμπληρώνει την ε, δημόσια και επαγγελματική σύνταξη. Οι συμπληρωματικές συντάξεις αποτελεσματικές μπορούν να είναι μόνο εάν είναι προσβάσιμες σε κάθε τάξη εισοδήματο. Σε κάθε κατηγορία εισοδήματο. Άρα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά και με ισχυρή απόδοση σε σχέση με το κόστος, έτσι ώστε να είναι ελκυστικά τα προϊόντα αυτά για όλους τους αποταμιευτές. Πρέπει να προσφέρονται λοιπόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα σύστημα ενιαία καταχώρησης ώστε να μην υπάρχει και επιπλέον να μην υπάρχει διασυνοριακός ανταγωνισμός μεταξύ των συστημάτων. Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λένε ότι θα πρέπει τα φορολογικά ε, κίνητρα να είναι αντίστοιχα με αυτά των συστημάτων που ήδη υφίστανται, ε, ακόμα και αν δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά τα PEPS ε με τα εθνικά συστήματα. Η αξιοπιστία του ΠΕΠ ε και ο ρόλος της ΑΕΟΠΑ δυστυχώς αποδυναμώθηκαν στη διαδικασία των τροπολογιών. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό το βήμα αυτό που πραγματοποιείται για την εισαγωγή μιας γνήσιας αγοράς ατομικών στεξιωτικών προϊόντων και έτσι ενισχύεται η κεφαλαιαγορά αγορά της Ευρώπης συνολικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις αλλά και ανάπτυξη και θέσεις εργασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα. Πολλή δουλειά έχει να γίνει ακόμα, μένει να γίνει ακόμα για να προσδιοριστούν κάποια επιμέρους σημεία των ΠΕΠΣ e με κατεξότηση πράξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και παρακολουθεί με προσοχή το έργο της ΑΙΟΠΑ ώστε να βεβαιώνεται πάντα πως οι κατεξοδοτήσεις συμπράξεις ακολουθούν πιστά τις ε, πολιτικές κατευθύνσεις που έχουν ορίσει οι συνομοθέτες. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Ο κύριος Μπέκερ, εκ μέρους της Επιτροπής Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ήμουν από εκείνου που αγωνίστηκαν υπέρ των ΠΕΠ εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία για ένα τέτοιο προϊόν, νέο θετικό για την νεότερη γενιά της Ευρώπης, γιατί εξασφαλίζει μια πρόσθετη σύνταξη με καλύτερη ποιότητα ζωής δηλαδή που θα προσφέρεται στην ε, προχωρημένη ηλικία. Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης ή σε άλλες περιοχές της Ευρώπης δεν υπάρχουν καλά ανεπτυγμένα συστήματα, αντίστοιχα δηλαδή με αυτά της ε, πατρίδας μου της Γερμανίας. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να εξασφαλίσει σαν λειτουργία το ΠΕΠ, δηλαδή και πρόσθετη αξία, προστιθέμενη αξία για βελτίωση και εξασφάλιση ενός επίπεδου ζωής στην ε, προχωρημένη ηλικία στην εποχή της σύνταξης. Ε, υπάρχουν διαφορές εναλλακτικέ που προσφέρονται, ιδιαίτερα το θεωρώ ότι υπάρχει μία βασική εκδοχή, πανευρωπαϊκή, ομοιόμορφη, με εγγυημένο κεφάλαιο επιπλέον που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για πολλούς πολίτες εκεί όπου δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένα τα σταξιωτικά συστήματα. Είναι ένα σύστημα διαφανές, ελκυστικό, και συμπληρωματικό στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα τη σύνταξη. Και ιδιαίτερα υπογραμμίζω αυτά που είπε η συγγήτρια κυρία Ινετφέλτ, ότι δεν είναι επουδενή ανταγωνιστικό προ τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα των συνταξιδοτικών συστημάτων, αλλά συμπληρωματικό και ω εκ τούτου προσφέρει πολύτιμη συμβολή στην διασφάλιση ε, των συνταξιδοτικών εισοδημάτων. Υπάρχει επίση μια τυποποιημένη τεκμηρίωση που θα πρέπει, προβλέπεται μάλλον μια τεκμηρίωση που θα πρέπει να προσφέρεται στον ε, πελάτη από τα μια Ε, από αυτήν θα εξαρτάται και η πιστοποίηση με την εγγύηση της ΙΟΠΑ και έτσι είμαι πεπισμένος πως προσφέρουμε στη νέα γενεά ένα εξαιρετικό σταξιδοτικό πρόσθετο προϊόν. Ευχαριστώ από πλευρά της αγοράς ΙΜΚΟ. Στάλφος Λάγγεν επίσης δύο λεπτά. Κόλιν Λάγγεν κυρία Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό κατά την τρέχουσα θητεία. Ω εισηγήτρια στην ΙΜΚΟ, καταρχά θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Ινφελτ. Την ευχαριστώ για την ε, καλή και ειλικρινή συνεργασία. Για μένα από την αρχή ο στόχος ε, αυτού του προϊόντος ήταν να είναι απλό, ασφαλές, διαφανές, φιλικό προς το καναλωτή, φτηνό και μακροπρόθεσμο προϊόν σύνταξη σύνταξης γύρατος. Και καταφέραμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Μετά την ολοκλήρωση των πραγματεύσεων, μπορώ να πω συνοψίζοντας, ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι κατάλληλη για νοστιργή αγορά και ε, χρήσιμη για τον καταναλωτή. Έτσι τη διαμορφώσαμε. Και το βασικό είναι να υπάρχει ένα βασικό ΠΕΠ. Κάθε ε, ένας που συμμετέχει στην αγορά θα πρέπει να προσφέρει τέτοιο βασικό ΠΕΠ και μάλιστα και ψηφιακά που να μπορεί φτηνά και ασφαλώς να συναυθεί. Και ε, το βασικό είναι η προστασία του κεφαλαίου για μένα. Το κεφάλαιο ενός βασικού ΠΕΠ δεν μπορεί ποτέ να χαθεί κατά τη γνώμη μου και δεν θα πρέπει να το ροκανίζουν ε, τα διάφορα στοιχεία του κόστους. Πρέπει λοιπόν αυτό να γίνεται μέσω εγγύησης του κεφαλαίου ή με τεχνικές μείωση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, του κινδύνου. Είναι ένα προϊόν συνταξιοδότης. Και αυτό μπορούμε να το ε, ε, διασφαλίσουμε ούτω ώστε να ένα 35% να ε, είναι εγγυημένη σύνταξη. Και προϋπόθεση για να επιτύχει είναι η στήριξη από τα κράτη-μέλη. Μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να ευνοήσουν με τον ίδιο τρόπο τα ΠΕΠ με διάφορα ε, παρόμοια εθνικά προϊόντα. Γι' αυτό χαιρετίζω τις τροπολογίες όπου λέει ότι οι προϋποθέσεις για το ΠΕΠ δεν θα πρέπει να είναι πιο ακριβές από τα εθνικά προϊόντα. Έτσι ολοκληρώνουμε ε, την ενιαία αγορά και βοηθάμε ιδιαίτερα τους νέους και τα άτομα με χαμηλό εισόδημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι ομιλητέ από πλευρά των ομάδων. Πρώτα απ' όλα ο κύριο Hayes για το ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Σοφή και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα σήμερα και ευχαριστώ και την Κομισιόν. Πέρσι στην Ιρλανδία 30.000 πολίτες ήρθαν να δουλέψουν γιατί έχουμε πλήρη απασχόληση στην Ιρλανδία. Πολλοί είναι νέοι. Πολλοί ήρθαν στην Ιρλανδία για να εργαστούν για 4-5 χρόνια ίσως και να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να αποταμιεύουν νωρίτερα, όπω είπε και ο επίτροπο, Και ένα από τα πλεονεκτήματα του ΠΕΠ είναι ότι έχουμε ένα πανευρωπαϊκό προϊόν. Δεν είναι το τέλο του ΠΕΠ, είναι το πρώτο βήμα. Κάνουμε πολύ μικρά βήματα εδώ σήμερα, αλλά είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για να στείλουμε το μήνυμα στου νέου που ταξιδεύουν στην Ιρλανδία και αλλού για δουλειά, να έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν ένα πανευρωπαϊκό συνταξιδοτικό προϊόν. Δεύτερο σημαντικό ότι αυτό αποτελεί τμήμα τη ε, κεφαλαγορά. Θα πρέπει να έχουμε τη σύνδεση μεταξύ των επενδύσεων ε, και των αποταμιευτών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται αυτό το προϊόν από πολλαπλού παρόχου. Έτσι λοιπόν, ο κλάδο ε, των ασφαλιστών και οι διαχειριστέ περιουσιακών στοιχείων μπορούν να παρέχουν τώρα αυτό το προϊόν σε πανευρωπαϊκή δάση αλλά θέλω να επαναλάβω ότι αυτό είναι ένα προϊόν τρίτου πυλώνα. Είναι ένα εκούσιο προϊόν, με κανένα τρόπο δεν υποσκάπτει τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα στι συντάξει. Αυτό είναι ένα προϊόν που βασίζεται στην προστασία των καταναλωτών, δίνει πλήρη διαφάνεια στους πολίτες για το κόστος και διασφαλίζει υποχρεωτική παροχή συμβουλών, έχει ισχυρέ συμβατικέ απαιτήσει, φορητότητα, όριο στην ε, στο τέλος και εποπτεία από τις αρμόδιε αρχές και την ΕΙΟΠΑ. Κάναμε μια καλή αρχή με την πρόταση αυτή. Δεν είναι το τέλος βέβαια τη υπόθεση αυτής κατά κανένα τρόπο, αλλά αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα στην Ευρώπη θα πρέπει να προβλέψουμε ότι μέχρι το 2060 θα έχουμε έναν εργαζόμενο για ε, δύο συνταξιούχους και αν δεν θέλουμε τους ανθρώπους να αποταμιεύσουν θα χειροτερεύει η κατάσταση με τα χρόνια. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Γκίγκολτ. Συμφωνείτε. Ο κύριος Γκίγκολτ. Thank for... Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε. Καταρχήν, θα πρέπει να δηλώσω ότι μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με τον Μπράιαν, πάντοτε σας συμπαθούσα ακόμη και αν συμφωνούσαμε σε πάρα πολλά θέματα. Ωστόσο, να πω ότι ο κώδικας διοντολογίας μας λέει στο σημείο 3.3 ότι πριν ε, να πάρει κανείς το λόγο, οποιοδήποτε δυνατή σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει γραπτός ε, ή προφορικός να δηλώνεται στον πρόεδρο. Δυστυχώς δεκτήκατε να εγκατέλειψετε τον οικό για να γίνετε διευθύνων σύμβουλος της Ιρλανδικής Τράπεζας. Έχετε δηλώσει ε, αυτή την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων όταν ασχοληθήκατε με το φάκελο αυτό. Ναι, το έχω δηλώσει, είναι η απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστέ, η κυρία Γιάκον Σάρη. Ένα λεπτό. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει μια πιο επικριτική στάση απέναντι στην πρόταση αυτή από ότι οι προηγούμενοι ομιλητές. Εγώ προσωπικά ήμουν αρκετά ενθουσιώδης. Εμείς ε, θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό που θέλουμε είναι να λειτουργήσει η ενιαία αγορά, να αυξηθεί η κινητικότητα των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν είναι κάτι που προωθεί την κινητικότητα και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αυτό πω αυτό που επικρίνουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή, αυτό που περισσότερο φοβούνται ως προς το μέλλον τους, είναι πως ε, όταν έχουν ε, ήδη εργαστεί κάποια χρόνια σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το συνταξιδοτικό σύστημα να μην ακολουθεί αυτή την κατάσταση. Και αυτό το προϊόν ΠΕΠ ουσιαστικά προκάλεσε κάποιους φόβους ότι πρόκειται για αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας. Όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών εμείς βελτιώσαμε πολύ το κείμενο και τώρα είναι σημαντικό να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και του κεφαλαίου τους. Αν προσελκύσει τον κόσμο αυτό το προϊόν, είναι γιατί πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο θα φέρει μια ευρωπαϊκή ετικέτα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ, ο κύριος Λουκ, ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η σύνταξη είχε πει κάποτε ο Νόρμπερτ Πλουμ, υπουργό εργασία τότε. Τώρα όμω δεν είναι τίποτε σίγουρο, ούτε καν η σύνταξη. Ούτε η χρηματοδότησή της, ούτε η ε, κεφαλαϊκού τύπου σύνταξη μπορεί να είναι σίγουρη. Και αυτό οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς δεν υπάρχουν πλέον επιτόκια που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της αποταμίευσης και άρα δεν μπορεί να υπάρχει κεφαλαιακή σύνταξη. Τεράστιο σφάρμα αυτό της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής μας Τράπεζας, το οποίο ούτε το ΠΕΠ μπορεί να ανατρέψει. Πολύ ωραία τα κίνητρα για την αποταμίευση. Όταν όμως δεν υπάρχουν επιτόκια, είναι μηδενικό ή ελάχιστο, ελάχιστη η απόδοσή τους. Είναι πολύ μικρό αυτό το οποίο μπορεί το Κοινοβούλιο με την πρότασή του να συμβάλλει προκειμένου να τρέψει αυτή την καταστροφική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάλι είναι επιπλέον πολύ περίπλοκο, αδιαφανές αλλά και πολύ ακριβό αυτό το προϊόν για την αγορά και έτσι δεν μπορεί να αποβεί αποτελεσματικό και επιτυχές. Διανοηθείτε ότι επιβάλλεται υποχρεωτική ενημέρωση και παροχή συμβουλών στον πελάτη, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου ικανός να την αντιληφθεί. Έτσι λοιπόν, ο πολιτής αυτών των προϊόντων ο πολιτή συγγνώμη των προϊόντων αυτών, ο οποίο αναλαμβάνει να, κάνει, να δώσει τι συμβουλέ αυτέ, είναι ανίκανο, δεν μπορεί να, τις, το εξηγήσει το προϊόν αυτό ικανοποιητικά. Ένα προϊόν που, όπω είπα, είναι ακριβό και αδιαφανέ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Γκίκολτ που επισήμανε διάφορα από αυτά στοιχεία. Ευχαριστώ, Καλβέτ Σαμπον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές και όσους βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του κειμένου. Πρόκειται για ένα θέμα τεχνικό και πολύπλοκο που συζητούμε εδώ σήμερα. Και όπως φαίνεται μπορούμε να φτάσουμε να μιλάμε και για τα λάθη στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Αυτό έχει τη φιλοδοξία που έχει. Και η φιλοδοξία που έχει, όπως ε, είπε από την πρώτη μέρα, ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Απασχόλησης είναι να διευκολύνει και να αυξήσει τις δυνατότητες για μια αξιοπρεπή σύνταξη για τα άτομα που για ιστορικούς ε, λόγους δεν μπόρεσαν ε, να έχουν ε, μια επαρκή κάλυψη στο δημοσιο σύστημα της χώρας τους ή έχουν υπερβολικά χαμηλή σύνταξη. Και επομένως είναι ένα ε, θέμα να θέλει να μπει η Ευρώπη και να προστατεύσει καλύτερα τους ηλικιωμένου μας. Συζητάμε για το αν είναι επαρκή ή εγγύης θεφαλαίου. Εντάξει, μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Η παρουσία της Ευρώπης ε, αρκεί με την ΕΙΟΠΑ. Θα θέλαμε κάτι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θετικό εργαλείο κοινωνικά και ε, είναι αστείο το να λέει κανείς ότι αυτό επιτίθεται στα δημόσια συστήματα, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι μια άχρηστη δημαγωγία. Από πλευρά της ΓΚΟΕ. Ένα λεπτό, ο κύριος Σίοντεμαν. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Χρειαζόμαστε ισχυρά συστήματα συνταξιοδοτικά και καλούς μισθούς για να έχουμε καλή δημόσια σύνταξη. Η ιδιωτικοποίησή της, όπως απέδειξε και μία έκθεση που δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ΠΕΠ, ε, αυτό καλεί να ενισχυθούν οι, οι δημόσιες συντάξεις και να σταματήσουν οι ιδιωτικές. Όχι μόνο είναι πολιτικά λάθος, αλλά είναι και κακοφτιαγμένο. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τους αγοραστές ότι αυτό το οποίο πληρώνουν τελικά θα το λάβουν ως εισόδημα. Είναι πολύ υψηλό το κόστος και υπεύθυνοι για τη χρήση του ΠΕΠ θα είναι αυτοί οι διαχειριστές των ΠΕΠ, ε, των hedge funds. Το 20% των εργαζομένων μας που απειλούνται από φτώχεια δεν πρόκειται να βοηθηθούν γιατί η σύνδεση με τις κεφαλαγορές είναι οπωσδήποτε επικίνδυνη και γι' αυτό εμείς απορρίπτουμε αυτό το ΠΕΠ και έχουμε κάνει τροπολογία να απορριφθεί. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Ο κύριος Άικχουτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την θαυμάσια εργασία της. Και ίσως το πιο σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ήδη υπάρχουν ιδιωτικά συνταξιωτικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά υπάρχουν χωρίς να υπάρχουν επαρκείς ρυθμίσεις. Αυτό που κάνουμε είναι επιτέλους να δημιουργούμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά σταξιωτικά προϊόντα. Και το καλύτερο σε αυτή την πρόταση είναι ότι δημιουργούμε ένα βασικό πανευρωπαϊκό ιδιωτικό συνταξιδοτικό προϊόν. Έχει κανόνες για να προστατεύονται οι καταναλωτές. Και δεν πρόκειται όχι να το αναλάβουν όλοι οι διαχειριστές υπεύθυνοι των hedge funds. Μπορείτε να επικρίνετε βέβαια αλλά υπάρχει και ένα το όριο για το σύνολο του κόστους του προϊόντος. Και η ερώτηση προς την Κομισιόν είναι, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το κόστος θα πρέπει να είναι το πολύ 1% του συνολικού κόστους. Αυτό είναι πολύ σημαντική διευκρίνηση. Τέλος, όλοι ξέρουμε ότι δεν αντικαθιστά τη βασική δημόσια σύνταξη, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πει σαφέστατα ότι δεν προωθούν περαιτέρω περικοπές του πρώτου πυλώνα. Δεν είναι θέμα λιτότητας. Θα είναι συμπληρωματικός αυτό, συμπληρωματικό αυτό το μέτρο τρίτου πυλώνα. Δεν θα αντικαθιστά. Ευχαριστώ. ΕΝΕΦ, e ο κύριος Ζούλστρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο αντιτάσσεται στα ΠΕΠ προϊόντα τα οποία θα οδηγήσουν σε εκβάθρον αναθεώρηση της νομοθεσίας των κατοχωρών έτσι και κατεψήφισε η Ολλανδή υπουργό στο Συμβούλιο την πρόταση αλλά με, με την αρχή της πλειοψηφίας βρεθήκαμε στη μειοψηφία. Ωστόσο, είναι σαφές ότι δεν επιτρέπεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να ε, επιβάλλει ρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα στα κράτη-μέλη. Έχω υποβάλει ερώτηση, απάντηση όμως δεν έχω λάβει ακόμα, ύστερα από δύο μήνες, και ρωτώ γιατί διαμορφώνονται αυτές οι πλειοψηφίες πάντα εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε μια χώρα όπως η δική μας που το σύστημα δουλεύει τόσο καλά και που άλλωστε και οι ομοσπονδίες των στεξούχων των κατοχωρών συμφωνούν σε αυτό γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια υπονόμευσης του συστήματός μας. γιατί το εθνικό μας σύστημα το οποίο δουλεύει τόσο καλά πρέπει να υπονομευθεί, γιατί πρέπει να χάνεται αυτή η κυριαρχία των κρατών μελών και όταν μάλιστα τα συστήματα της εξωτικά δουλεύουν τόσο καλά. Είναι πολύ ωραίο βεβαίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν ε, βιώσιμα συστήματα συντοξιωτικά αλλά ένας λόγος παραπάνω, να μην μπλέκεται και να μην τα καταστρέφει. Υπάρχουν πολλές, πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στη νέα πρόταση. Ξέρουμε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε ένα ζήτημα και παραβιάζει τι αρχές τη εθνική κυριαρχία και καταστρέφει τα εθνικά συστήματα. Θα καταψηφίσουμε βέβαια. Η πρόεδρο, ο κύριο Ζαριανόπουλο, μία εγγεγραμμένο, έχετε ένα λεπτό. Το πανευρωπαϊκό ατομικό ασφαλιστικό προϊόν που αποφασίζεται σήμερα είναι πανευρωπαϊκή ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση κίνδυνος θάνατος για τους εργαζόμενους ιδιαίτερα τους νέους. ένα μεγάλο εμπόδιο στην κερδοφορία ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου οι κατακτήσεις δηλαδή σε συντάξεις και υγεία η δημόσια κοινωνική ασφάλιση μετά από χρόνια περικοπών ισοπεδώνονται. Επιχειρήσει και κράτο όχι μόνο απαλλάσσονται από το βάρο του, αλλά κερδοσκοπούν στι πλάτε των εργαζόμενων. είναι καθαρή ιδιωτική ασφάλιση συμπλήρωμα σε κρατικέ συντάξει πείνα για δουλειά ω θανάτου με ενεργό γύρανση αν βέβαια σου μένουν για να επενδύσει με τσακισμένου μισθού. Καμιά απολύτω εγγύηση ότι θα πάρει πίσω όσα έδωσε. Όλα τα αποθεματικά στο τζόγο των χρηματιστηρίων, τζάμπα χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα ακόμα δώρο σε αυτέ τι τράπεζε και τι ιδιωτικέ ασφαλιστικέ συναγερμός τώρα για εργαζόμενους παλιούς και νέους μαύρο στο πραγματικό μέτωπο νεοφιλελεύθερων σοσιαλδημοκρατών δίθεν αριστερών τύπου σύριζα που κρύβουν την ταύτισή τους και εδώ με ψεύτικα δίπολα και διλήμματα. ταξικός αγώνας ενίσχυση των κομμουνιστών είναι η μόνη εγγύηση για κοινωνική ασφάλιση και εργατικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Περνούμε στους επόμενους ομιλητές, στους ομιλητές, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είμαι από εκείνου τους βουλευτές που υποστήριξαν αυτή την πρόταση. Την προσυπογράφω και θέλω να επισημάνω ότι φόβοι των συναδέλφων που υπονομεύονται τα εθνικά συστήματα ε, θεωρώ πως είναι αβάσιμοι. Έχει σημειωθεί επανειλημμένως ότι πρόκειται για ένα συμπληρωματικό προϊόν για τον πολίτη εκείνον που ρωτάτε πώς μπορεί να έχει περισσότερα εισοδήματα στην ε, ε, ηλικία της συνταξιοδότησης. Είναι καλό να υπάρχει ένα τέτοιο προϊόν, μια ακόμη επιλογή για τον πολίτη να αποταμιεύει εν ώψη των γυρατιών του. Ένα προϊόν λοιπόν τρίτου πυλώνα, ένα προϊόν το οποίο δεν υπονομεύει εμποδενή τα εθνικά συνταξιωτικά συστήματα. Είναι πράγματι Αβάσιμη η φόβη ορισμένων εκ των συναδέλφων, γιατί κανείς δεν μιλάει για ανατροπή ή για καταστροφή των εθνικών συστημάτων συνταξιδότησης και των ε, ιδιαιτεροτήτων τους. Ένα τέταρτο, 25% μόνο των συνταξιούχων έχουν ιδιωτικά συνταξιδοτικά προϊόντα και αυτό είναι πολύ μικρό ποσοστό. Η δουλειά, η γενιά των ενεργών σήμερα πολιτών, εκείνων που εργάζονται, δεν θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τις συντάξεις της από το κράτος. Δεν θα μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί τις συντάξεις τους. Άρα πρέπει να μάθουν αυτοί οι πολίτες ήδη από τώρα να αποταμιεύουν. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Θα ήθελα να επισημάνω πάντως ότι θα προτιμούσα το προϊόν αυτό να είναι πιο φιλόδοξο. Καλό θα ήταν να είχαν συμφωνήσει Συμβούλιο και Επιτροπή σε φορολογικά κίνητρα ε, ανταγωνιστικά έναντι των εθνικών προϊόντων, ώστε να είναι πιο ελκυστικό το προϊόν για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό ζήτημα, σήμερα στην Ευρώπη όταν μιλάμε για τις συντάξεις, περισσότερο μας ενδιαφέρει να μιλάμε για τον πρώτο πυλώνα. Δηλαδή, πώς θα εγγυηθούμε ότι ο καθένας στο τέλος της διαδρομίας του μπορεί να έχει μια ε, επαρκή σύνταξη. Τώρα, να μιλάμε για έναν ιδιωτικό συντοξιδικό πυλώνα, δηλαδή για τον τρίτο πυλώνα, σκεφτόμενοι ότι αυτό ο τρίτο πυλώνα θα μπορεί να λύσει το ζήτημα του πρώτου πυλώνα, νομίζω ότι είναι ε, κακή κατεύθυνση. Και μάλιστα όταν διαβάζουμε και τις συστάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συχνά στο πλαίσιο των συστάσεων διαβάζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη να μειώσουν τις δαπάνες τους ε, για το συνταξιδοτικό του πρώτου πυλώνα και βλέπουμε ότι η λογική θα ήταν να ε, μεταφερθεί προς τον τρίτο πυλώνα, προς τις ιδιωτικές συντάξεις. Δηλαδή η συζήτηση που έχουμε σήμερα μου φαίνεται πολύ ε, ιδιαίτερη γιατί οι προτεραιότητε μα θα έπρεπε να πάνε προ τον πρώτο πυλώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σημερινή πρόταση τη ιδιωτική συντάξη, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετέ δυσκολίε και μία κυρία δυσκολία είναι να πούμε ότι η φορητότητα μπορεί να γίνεται σε δύο κράτη-μέλη, ενώ ε, λέμε ότι βάζουμε μία ετικέτα πανευρωπαϊκού προϊόντο. Και το τελευταίο σχόλιο που έχω να κάνω αφορά το θέμα τη φοροδιαφυγή που μπορεί να ε, γίνει μέσω του ιδιωτικού πυλώνα συνταξιοδότηση. Δηλαδή, μπορεί να πληρώνουμε εισφορέ σε μια χώρα και να πάρουμε σύνταξη σε μια άλλη χώρα, επιλέγοντα τη χώρα που έχει τα περισσότερα φορολογικά ωφέλη. Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή η πρόταση που συζητούμε σήμερα δεν απαντά στην προβληματική των συντάξεων στην Ευρώπη σήμερα και μάλιστα ευνοεί το θέμα τη φοροαποφυγή σε ό,τι αφορά την κεφαλαιοποίηση. Δεν θα υπερψηφίσω λοιπόν την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Σταρμπάτη δεν είναι στην αίθουσα από ό,τι βλέπω. Παρακαλώ τον κύριο Σελίμωβιτς να λάβει το λόγο για ένα λεπτό και τριάντα δεύτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο θα κατορθώσει να ψηφίσει αυτό το σύστημα και θα βοηθήσει ε, τους Ευρωπαίους ε, να έχουν ένα τέτοιο συνταξιδοτικό προϊόν. Σήμερα ε, στην αγορά υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που πολλούνται, όμως ό,τι αφορά το κεφάλαιο έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Φέροντας αυτό το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιδοτικό προϊόν θα είναι πιο εύκολο να αποταμιεύσουν οι άνθρωποι και θα λάβουν σύνταξη σε μια χώρα όπου μπορεί σήμερα να μην είναι δυνατό να τη λάβουν και θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αν μετακινηθούν σε άλλα χώρα χωρί Νομίζω ότι αυτό είναι στι καλέ ειδήσει για του Ευρωπαίου πολίτε. Αν δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι υποχρεωτικό το σύστημα, είναι κούσιο και δεν αντικαθιστά το εφιστάμενο σύστημα, απλώ ε, το συμπληρώνει. Και θα βοηθήσει και του παρόχου και του καταναλωτέ. Δεν βλέπω λοιπόν που είναι το πρόβλημα. Ξέρω ότι χρειάστηκαν δεκαετίες ε, σχεδόν ε, για να υλοποιηθεί και ξέρω ότι υπήρχε αντίσταση και από την χρηματοοικονομικό κλάδο ε, σε κάποιες χώρες. Όμως για μένα αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ωφελεί τον ανταγωνισμό και έχει και θετικές συνέπειες για τους πολίτες ουσιαστικά τι πετυχαίνει. Θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες που δεν μπορούν να έχουν αξιοπρεπή συντάξει σε κάποιες χώρες σήμερα να τις λάβουν. Θα είναι πιο φορητό, ευκολό κατανοητό προϊόν και σίγουρα θα είναι πιο φτηνό για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και για τους πολίτες τους. Αυτό μπορεί να κάνει η αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Σας ευχαριστώ κυρία έχω Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε υπό το μύθο ότι εσείς οι ίδιοι έχετε δημιουργήσει μη βιωσιμότητα στις δημοσίες συντάξεις, προωθείτε ένα προϊόν που ανοίγει ένα νέο μέτωπο για την κερδοσκοπία στην Ευρώπη, ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που ποτέ δεν θα μπορέσει να αντικαταστεί, να αποτελήσει καμία εγγύηση για τους πολίτες και ωφελεί μόνο μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων τους πιο πλούσιους ε, και τις τράπεζες. Ουσιαστικά διοχετεύει τις αποταμιεύσεις των πολιτών στι χρηματαγορέ. Εσεί μόνο θέλετε να διευρύνετε την ενιαία αγορά κεφαλαίων με γιγάντια συνταξιδοτικά ταμεία που θα μπορούν να παρεμβαίνουν στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Το καθήκον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών θα έπρεπε να είναι να προστατεύσουν του πολίτε. και εσεί δεν σέβεστε αυτή την αρχή ενισχύοντα ιδιωτικά συστήματα υψηλού κινδύνου που ούτε καν έχουν αγγίσει κεφαλαίου πραγματικού όρου. Θέλετε πράγματι προστατεύσετε τους πολίτες. Η μόνη οδός είναι να ενισχύσετε τα δημόσια συνταξιδοτικά συστήματα που είναι ο μόνος και ο μεγαλύτερος μηχανισμός καταπολέμησης της στόχης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γκίκολτ, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα πολύ αντιφατικά επιχειρήματα κατά αυτού του συνταξιωτικού προϊόντος. Είναι απόλυτα σαφές ότι η βάση των συντάξεων πρέπει να είναι οι δημόσιες ε, συντάξεις και δεν πρόκειται αυτό το προϊόν να έχει χρηματολογικά, συγγνώμη, ε, φορολογικά πλεονεκτήματα. Και αυτό είναι σωστό, διότι κυρίως πρέπει να επικεντρώνουμε στις δημόσιες συντάξεις. Όμως, Ούτως ή άλλως υπάρχει πάρα πολύ σπέκουλα με τα ιδιωτικά στα εξωτικά προϊόντα και αυτό το κείμενο θα περιορίσει αυτή τη σπέκουλα και αυτό ακριβώς είναι πλεονέκτημα για τους εργαζόμενους και τους ηλικιωμένους που δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να επιλέξουν τα καλύτερα προϊόντα στην ιδιωτική αγορά και δεν έχει τίποτα να κάνει με την ε, φοροδιαφυγή. Διότι εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σύνταξη σε μια χώρα και μετακομίσει αλλού, αυτό δεν είναι φοροδιαφυγή. Αυτό είναι η ελεύθερη επιλογή τόπου διαμονής. Θεωρώ ότι πολλοί τα μπερδεύουν όλα για να κατηγορήσουν αυτό το προϊόν. Κύριε Γκίγκολτ, η κυρία Αβενά έχει ζητήσει μία μπλε κάρτα. Συμφωνείτε. Παρακαλώ, κυρία Αβενά. Ευχαριστώ. Κύριε Γκίγκολτ, όταν λέτε οι άνθρωποι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, όταν κερδίσει κανείς 1200 ευρώ το μήνα, νομίζετε ότι μπορείτε να πληρώσετε ιδιωτική ε, σύνταξη για να έχετε περισσότεροι στα 65, λέτε ότι δεν θα υπάρξει φοροδιαφυγή. Αλλά γι' αυτό εμείς ζητήσαμε σε αυτή τη διαδικασία η σύνταξη όταν είναι προϊόν κεφαλαιοποίησης να ε, σας χορηγείτε στη χώρα όπου έχετε πληρώσει τις συνεισφορές σας. Και δεν το επιτύχαμε. Δηλαδή όταν θα βγείτε από αυτό το συνταξιδοτικό ταμείο θα πάτε να το κάνετε αυτό στη χώρα που σας ωφελεί περισσότερο φορολογικά. Το επιχείρημά σας είναι επιχείρημα για τους πλούσιους και δεν έχει έννοια. Ναι, ναι, τα είπαν πολύ δυνατά αυτά, αλλά πρέπει να πω στην πραγματικότητα η κατάσταση έχει ως εξή. Πρώτα, για μένα το να είναι κανείς φτωχός ε, και εργαζόμενος που δεν βγάζει πολλά ε, αρχίζει από χαμηλότερη ε, αμοιβή από τα 1200. Όμως γιατί κάποιοι μπορούν να αποταμιεύσουν μικρά ποσά και θα, μπορούν, θα έπρεπε να μπορούν να τα αξιοποιούν. Η, επιχειρημα, η, η επιχειρηματολογία σας είναι εθνικισμός των συντάξεων. Δηλαδή, αν έχετε πληρώσει για σύνταξη σε μία χώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να μείνετε εκεί. Εγώ το θεωρώ είναι πολύ φυσιολογικό ένα Γάλλο να πάει στην Ισπανία να ζήσει όταν πάρει σύνταξη. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Και αν το σύστημα είναι διαφορετικό στην Ισπανία, είναι διαφορετικό. Αλλά αυτό σημαίνει ελευθερία στην Ευρώπη. Παρακαλώ, εσεί για ένα λεπτό. Πρέπει να είναι ο σεβασμό των πολιτών και του κόπου τη εργασία του. Επιδίωξή μα, ο περιορισμό τη ιδιωτικοποίηση και η ενίσχυση των δημόσιων καθολικών συστημάτων κοινωνική ασφάλιση. Εν προωθείται ένα αμυγό επενδυτική φύσεω προϊόν υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη το οποίο μάλιστα θα χαίρει φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων. οι αρχέ ενό δίκαιου και βιώσιμου συστήματο είναι απλέ υποχρεωτική ασφάλιση εγγυημένη επαρκή σύνταξη αναλογικότητα και σταθερότητα των εισφορών ανταποδοτικότητα παροχών υποστήριξη της συνέχεια των εισφορών με όρους αναδιανομής μακροχρόνια δομημένη αποταμίευση και δημιουργία αποθεματικών ώστε το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα να είναι βιώσιμο και αξιοπρεπέ για του πολίτε. βέβαια κάθε πολίτη πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει τυχόν επιπρόσθετε ιδιωτικέ συνταξιοδοτικέ επιλογέ. Όμω, και συνταξιοδοτικές επιλογέ. Όμω, η πολιτεία έχει την ουσιαστική υποχρέωση να καθορίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο με κατάλληλου κανόνε ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία του ανταγωνισμού ει βάρο του κρατικού συστήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπενιφέη, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η σημερινή ψηφοφορία σήμερα στην Ολομέλεια για το Πανευρωπαϊκό ατομικό εξωτικό προϊόν του τρίτου πυλώνα που θα είναι συμπληρωματικό στις ε, δημόσιε συντάξει έχει τεράστια σημασία. Μπορεί το ΠΕΠ λοιπόν να προσφέρει δυνατότητες για ενίσχυση της ατομικής ε, αποταμίευσης, να συμπληρώνει τη σύνταξη, να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, να βοηθήσει στην ενοποίηση των αγορών κεφαλαίων κατά τρόπο συγκεκριμένο. Βεβαίω το ΠΕΠ μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο αντιμετωπίζοντας ε, το μεγάλο χάσμα στα επίπεδα συντάξεων που γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των κρατών μελών. Βεβαίως θα είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικά, ελκυστικά για το κοινό. Καλό θα είναι να εγκαθιδρυθεί επιτέλους ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για τους νέους εκείνους που ζουν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όχι στις χώρες προέλευσής τους. Και έτσι μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα μοναδικό συνταξιδοτικό σπληρωματικό προϊόν που θα υπολογίζει διαφορετικές περιόδους ε, εργατικών εισφορών στα κράτη-μέλη, σε διάφορα κράτη-μέλη. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να υπάρχει εποπτεία στο σύστημα, στην διαχείριση των ε, εισφορών και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο μέλλον με τη λειτουργία του συστήματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Νάχτεγκαλ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκλέγομαι στην Ολλανδία από Ολλανδούς πολίτες. Χρειάστηκε λοιπόν να δοθεί και το αναγνωρίζω αυτό μια νέα όθηση στην ε, ε, στα εξωτερικά μας συστήματα. Ε, έχουμε ένα τεράστιο κεκτημένο εξωτικών συστημάτων 113 δισεκατομμύρια ευρώ στι κάτω χώρες έχουν αποταμιεύσει οι Ολλανδοί για τη ε, γυρατσιά τους. Το ίμιση του ενεργητικού των Ευρωπαϊκών Στατιωτικών Ταμείων το έχουν αποταμιεύσει οι ίδιοι οι Ολλανδοί. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται νέο στατιωτικό προϊόν και αντιτίθεμαι σε αυτό. Μόνο παρέμβαση σε ένα ε, εθνικό και επιτυχημένο προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σημάνει αυτό το προϊόν. Πρέπει οι ίδιοι οι Ολλανδοί να αποφασίσουν πώς θέλουν να οργανώσουν τη σύνταξή τους. Ευχαριστώ, Ουρμπαν Κρέσπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε οι συνταξιούχοι έχουν βαρεθεί να ακούνε τα θεσμικά όργανα να λένε ότι τα δημόσια συνταξιδικά συστήματα δεν είναι βιώσιμα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν εργαστεί όλη τους τη ζωή για να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη και ως κοινωνία υποχρεούμαστε να εγγυθούμε τις συντάξεις τους. Δεν είναι ένα θέμα κερδών αλλά δικαιωμάτων. Οι συνταξιούχοι δεν ε, χρειάζονται να παίζουν το καζίνο κανείς με τις συντάξεις τους ούτε να εφευρεθούν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα που το μόνο που το επιτρέπεται είναι να εμπορεύονται τι αποταμιεύσει του. Αυτό που χρειάζονται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί κάθετα στο να εγγυηθεί τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα και να σταματήσει να προωθεί την ιδιωτικοποίησή τους ε, και από εδώ προσφέρουμε όλη μας την υποστήριξη σε συνταξιούχους ε, που αγωνίζονται και εργάζονται και δείχνουν και υπερασπίζουν ε, τα δικαιώματα όλων, όχι μόνο τα δικά τους δικαιώματα, αλλά όλων τα δικαιώματα. Ας υπερασπίσουμε τις δημόσιες συντάξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ένα λεπτό κυρία Μιράντα. Αυτή την ε, εβδομάδα οι ευρωβουλευτές ε, λάβαμε πάνω από 20.000 ε, mail από τους συνταξιούχους που μας ζήτησαν να καταψηφίσουμε την πρόταση αυτή αξιοπρεπείς συντάξει, γιατί ένας άνθρωπος που λαμβάνει μια σύνταξη 400 ευρώ ή 600 ευρώ ή 700 ευρώ όπω πολλές φορές συμβαίνει στη δική μου χώρα είναι πολύ δύσκολο να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο προϊόν κύριε Επίτροπε. Επίση, το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει φορολογικές αρμοδιότητες έτσι λοιπόν κρύβεται εδώ μια παγίδα γιατί αφού έχουμε πάρα πολλές περικοπές ε, ε λόγω των αποφάσεων της ε, Τρόικας ε, και των διάφορων μεταρρυθμίσεων που είχαμε στο συνταξιδοτικό που προηθήθηκαν από το Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία, οι συνταξιούχοι μα ε, βλέπουν ε, ακροτεριασμένα τα δικαιώματά του και δεν ξέρουμε αν οι μελλοντικέ γενιέ θα λάβουν σύνταξη. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το προϊόν ε, τελικά του πιο πλούσιου θα ωφελήσει και θα χρησιμοποιήσει κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού, όπω η δημιουργία θέσεων εργασία και η βοήθεια στου λιγότερο ευνόμενου. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δηλώσω την υποστήριξή μου εδώ στου συνταξιούχου. Ευχαριστώ κύριο Στάνγκ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ένωση Κεφαλαγορών που ξεκίνησε κατά την τρέχουσα θητεία είδαμε δεκάδες προτάσεων αλλά δεν ξέρω πόσο βοηθάνε προτάσεις όπως το ΠΕΠ την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Οι προτάσει αυτέ δεν προωθούνται. Την επόμενη θητεία θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολλέ προσπάθειε για να βελτιωθεί αυτή η πρόταση. Αλλά γιατί είναι πανευρωπαϊκό αυτό το προϊόν, εάν η επίβλεψή του θα πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα συνολικά για τι προτάσει για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Και τι εννοείται θελούσιο προϊόν. Πώ θα συμβάλλει στο ε, σύστημα συντάξεων στις χώρες όπου δεν είναι επαρκές. Και γιατί θα πρέπει να ενδιαφερόμεθα για ένα τέτοιο προϊόν. Αυτό επειδή είναι τόσο χαμηλά τα επιτόκια βεβαίως. Στην Ολλανδία η στάση μας είναι ότι εντάξει ε, δεν θα κάνει κακό αλλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστή προσέγγιση προς την νομοθεσία γι' αυτό νομίζω πρέπει να το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε διαδικασία Catch the Eye. Τρεις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μαρίνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω από την αρχή ότι αφού άκουσα όσα υπόθηκαν εδώ από τα διάφορα μέρη, εγώ θα υπερψηφίσω την πρόταση αυτή. Γιατί θεωρώ ότι δεν ε, θα ανταγωνιστεί τα εθνικά συστήματα, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν αποταμιεύσει να μπορούν να μπουν σε ένα νέο συμπληρωματικό σύστημα, το οποίο δεν είναι ανταγωνιστικό με τα εθνικά συστήματα. Συμπληρωματικό θα είναι. Αυτό δεν είναι για όλους, ούτε καν αμφισβητεί τα εθνικά συστήματα, τα οποία θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με ένα καθολικό υποχρεωτικό μοντέλο για όλους ε, αυτό αφορά τα άτομα που τώρα αποταμιεύουν κατά κάποιο τρόπο και θέλουν να επενδύσουν αυτές τις ε, αποταμιεύσεις ε, τώρα μπορούν να επενδύσουν καλύτερα για το μέλλον τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή αυτή η πρόταση και ακριβώς σκοπεύει να συμπληρώσει και όχι να ανταγωνιστεί τα εθνικά συστήματα. Η κυρία Κούρεβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε λίγο πριν τις εκλογές τι μήνυμα θα στείλει το Ευρωκοινοβούλιο στους πολίτες ότι θέλει να κάνει στο τέλος της θητείας μας πιο πλούσιο τους μεγάλους παίκτες των αγορών με τις οικονομίες των εργαζομένων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βιάζεται να ενισχύσει τις αγορές με τις αποταμιεύσεις των εργαζομένων που αγωνιούν για τα κεράματά τους από την άλλη, οι κυβερνήσει δεν μπορούν να συμφωνήσουν καν για τα επιδόματα των εργαζομένων όταν μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Σας καλώ να αλογιστούμε και να δεσμευτούμε πώς θα ενισχύσουμε τη δημόσια σύνταξη καταψηφίζοντας την πανευρωπαϊκή ιδιωτική σύνταξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σέντρα Γοντρίγες. Μικρόφωνο παρακαλούμε για την ομιλήτρια. Μικρό. Α. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, συνάδελφοι. Εμένα αυτό το πανευρωπαϊκό τομικό συντοξιδοτικό προϊόν μου φαίνεται προσβλητικό απέναντι στους εργαζομένους, απέναντι στους επισφαλείς νέους, απέναντι στις γυναίκες, απέναντι σε τόσους ανθρώπους που δεν έχουν απασχόληση. Πιστεύω ότι για να εγγυηθούμε πράγματι δημόσια συνταξιδοτικά συστήματα και αξιοπρεπεί συντάξει, θα πρέπει να καταψηφίσουμε αυτό το πανευρωπαϊκό τομικό συνταξιδοτικό προϊόν και να εργαστούμε για τη θέσπιση μέτρων και ενό κανονισμού που πράγματι να βοηθήσει τα κράτη να ενισχύσουν τα δημόσια συνταξιδοτικά συστήματα προκειμένου να υπάρχουν αξιοπρεπεί συντάξει το μέλλον μας ε, δεν μπορεί να ε, εξαρτηθεί από την ικανότητα αποταμίευσης. Επίσης νομίζω ότι είναι έλλειψη ιδεοντολογίας να χρησιμοποιούμε δημόσια χρήματα ε, και να υποστηρίζουμε με φορολογικά κίνητρα αυτά τα ιδιωτικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο χρήμα δίνεται σε όσους θέλουν να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ κύριο Επίτροπος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη για την πολύ διαφωτιστική αλλά και κάπως έντονη συζήτηση για αυτό το σημαντικό θέμα. Καταρχάς, να διευκρινίσω, το πιο σημαντικό για όλους μας είναι τα δημόσια συνταξιωτικά συστήματα να είναι ανθεκτικά και να μπορούν να χορηγούν αυτό που πρέπει να χορηγήσουν σε πολλά κράτη-μέλη, αν όχι σε όλα, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η μεταρρύθμιση των δημοσίων ε, συνταξιδοτικών συστημάτων ούτως ώστε να είναι ανθεκτικά. Παρά το ότι αυξάνεται ο αριθμός ε, των ηλικιωμένων στις κοινωνίες μας. Αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχυθούν τα δημόσια συνταξιδοτικά συστήματα. Αυτό όμως το προϊόν, το ΠΕΠ, δεν έχει να κάνει με τα δημόσια σταξιοδοτικά συστήματα. Δεν τα αντικαθιστά. Απλώς προσφέρει περισσότερες εναλλακτικέ για τους πολίτες μας, τους απλούς πολίτες μας. Σε πολλά κράτη-μέλη. Αν δείτε τις στατιστικές θα δείτε ότι οι εργαζόμενοι που έχουν προσωρινές θέσεις εργασίας που δεν έχουν σταδιοδρομίες δεκαετιών που εργάζονται για σύντομα χρονικά διαστήματα και που θέλουν να συμπληρώσουν τις δημόσιες συντάξεις τους με ένα ιδιωτικό συνταξιωτικό προϊόν, τι μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή. Έχουν κάποιες δυνατότητες, αλλά τώρα δημιουργούμε κανόνες, ένα αριθμιστικό πλαίσιο για τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά συνταξιωτικά προϊόντα. Είναι λάθος αυτό, όχι δεν νομίζω. Αντίθετα, είναι θετικό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων ε, τέτοιων προϊόντων και συνήθω ε, οδηγεί σε πιο ασφαλή, ποιοτικά καλύτερα και φτηνότερα τέτοια προϊόντα για τους χρήστες. Ξέρω ότι ένα τέτοιο θέμα είναι πολύ εύκολο να αξιοποιηθεί για παραπληροφόρηση. Και για να αρχίσει η κινδυνολογία ότι ιδιωτικοποιείται η δημόσια σύνταξη. Μα δεν ισχύουν όλα αυτά. Κοιτάξτε, και τα τρόφιμα τα πουλάνε ιδιωτικέ εταιρείε. Τι θα έπρεπε να μην τα πουλάνε. Ξέρω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικέ ιδεολογίε και προτεραιότητε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί σε αυτή την αίθουσα που θέλει συνειδητά να παραπληροφορήσει του ψηφοφόρου γιατί δεν έχει έννοια, δεν είναι υπεύθυνο. Καλύτερα να εξηγήσετε τι σημαίνει πραγματικά αυτή η πρόταση, πώ θα βοηθήσει τις κοινωνίες μα. και παράλληλα βεβαίω, να στείλουμε το μήνυμα ότι όλοι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τι δημόσιε συντάξει στο μέλλον, που θα είναι λιγότεροι εργαζόμενοι και περισσότεροι συνταξιούχοι που θα πρέπει να αποφελούνται από αυτέ τι δημόσιε συντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε ή συγγετρία. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τους συναδέλφους εκείνους που υποστήριξαν στις ομιλίες τους και θα ήθελα ιδιαίτερος να αναφέρω τους και οδησηγητές και τις προεδρίες, ιδιαίτερος την Αυστριακή που συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς τους συναδέλφους ωστόσο οι οποίοι τοποθετήθηκαν πολύ αρνητικά και που σκοπεύουν να καταψηφίσουν την πρόταση εκ των οποίων μάλιστα οι περισσότεροι έχουν ήδη αποχωρήσει από το ημικύκλιο γιατί προφανώς δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν τα ε, σχόλια μας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλά fake news ακούστηκαν ότι δηλαδή, επί παραδείγματι, εάν κανείς το καταψηφίσει μπορεί να αποκλείσει από την αγορά την εισαγωγή αυτού του συστήματος. Όχι, του αντίον. Όποιος καταψηφίσει την πρόταση ενισχύει τους ε, καιροσκόπους, τους cowboys αυτής της αγοράς, γιατί ήδη υπάρχουν τα προϊόντα στην αγορά, εμείς απλώς τα πλησιώνουμε. Ή επίσης υπόθηκε ότι καταστρέφονται τα εθνικά στα εξωτικά συστήματα. Αιδίες, ανοησίες ήδη υπάρχουν και είναι απολύτως ανεξάρτητα αυτά. Καταψηφίζοντας ένα καλό κανονισμό ΠΕΠ e με προστασία του καταναλωτή, ουσιαστικά δεν κάνετε αυτό που θα έπρεπε να κάνετε, δηλαδή να στραφείτε προ τι εθνικέ σα κυβερνήσει και να του πείτε να συγυρίσουν τα εθνικά συντοξιδοτικά συστήματα και να τα τακτοποιήσουν έτσι ώστε να αποδίδουν καλύτερα. Για δε του Ολλανδού φίλου θα πρέπει να στραφώ, να, να αλλάξω και να μιλήσω, να αλλάξω γλώσσα και να μιλήσω Ολλανδικά. Για άλλη μια φορά λοιπόν ακούστηκε πω ε, σύνταξη στην Ευρώπη από του Ολλανδού ότι ε, όταν μιλούμε για σύνταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο συνταξιδοτικό σύστημα της, ε, των κατοχωρών. Ανοησίες, αηδίες, ανοησίες αγαπητοί συνάδελφοι και από τους φιλελεύθερους και από τους ελιστές και από, τους, ε, και από τις άλλες πλευρές. φοροδιαφυγή είπαν κάποιοι άλλοι. Μα ένα λεπτό δεν έχει καμία σχέση το ΠΕΠ με τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Δεν έχει καμία σχέση με φορολογική πολιτική το ΠΕΠ. Και δεν αλλάζει τίποτε στις φορολογικές πολιτικές. Είναι ανοησίες αυτά που διαδίδονται. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν κανονισμό που αποτελεί μια απόπειρα να δημιουργηθούν ε, προδιαγραφές προστασίας για προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά. Θα έπρεπε να μας συγχαίρετε, θα έπρεπε να επικροτείτε καθώς λάβαμε υπόψη και όλες τις τροπολογίες της ομάδας σας ε, που, των σοσιαλιστών δηλαδή που δεν ήταν και σύμφωνες με όλων παράδειγμα του κυρίου Γκουαλτιέρη. Άρα θα έπρεπε οι σοσιαλιστές να είναι ικανοποιημένοι. Μάλιστα βλέπω λέει η κυρία Πρόεδρος ότι ξεκινάει η προεκλογική εκστρατεία εδώ μέσα, ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση, η ψηφοφορία λαμβάνει λαμβάνει χώρα σήμερα το μεσημέρι και προχωρώ στην έκθεση Κάζα συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου για ε, γονείς και φροντιστές. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κάζα. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στην Ολομέλεια. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η οδηγία θα οδηγήσει στο να υπάρχουν επενδύσει στην οικογένεια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί ένα σωροπημένο νομοθέτημα που εισάγει ελάχιστες απαιτήσει που δίνοντας ε, πρόσβαση σε άνδρες και σε γυναίκες για γονική άδεια, άδεια πατρότητας και άδεια μέρημνας. Όπως επίσης και τη δυνατότητα να ζητήσουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Αυτή η οδηγία εισάγει άδεια 10 ε, ημερών για τους πατέρες, 2 ε, μήνες γονικής άδειας, 5 μέρες άδειας για τους φροντιστές και τη δυνατότητα οι γονείς να ζητήσουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Ο στόχος αυτής της οδηγίας πηγαίνει πολύ παραπέρα από το να προσθέτει δικαιώματα για τους γονείς και τους φροντιστές οδηγεί σε μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος επιμερισμός των ευθυνών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επέμενα πάντοτε ότι πρέπει να εξαλείψουμε την ανισότητα ε, των δύο φύλων ε, σε ό,τι αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωής. Ο στόχο μου είναι να το πετύχουμε αυτό έτσι ώστε ε, να ωφελούνται όχι μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες. Διάφορες μελέτες μας έδειξαν ότι παραδοσιακά οι γυναίκες είναι αυτές που αναλαμβάνουν περισσότερες ε, ευθύνες ε, για την ανατροφή των παιδιών. Όμως το αποτέλεσμα είναι θετικό για τους γονείς και τους φροντιστές και υπάρχει ε, ουσιαστικά επίπτωση και στις συντάξεις ε, και στους μισθούς. Γι' αυτό με αυτό το μέτρο θα είναι πιο εύκολο να μοιραστούν οι γονείς την ανατροφή των παιδιών ή να φροντίσουν τους συγγενείς τους. Αυτό θα διασφαλίσει ότι εμπλέκονται και οι άντρες ε, όσο και οι γυναίκες στο πρώτο χρόνια της ζωής των παιδιών τους. Επίσης θα υποστηριχτούν οι γυναίκες για να μπουν στην αγορά εργασίας χωρίς να αφαιρείται το δικαίωμα των παιδιών γονιών να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους. Οι γυναίκες θα λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη για να μπορούν να αναπτύξουν το δυναμικό τους στην αγορά εργασίας. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πατέρες ε, συμμετέχουν περισσότερο στην ανατροφή των παιδιών. Γι' αυτό πρέπει να παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να τους βοηθήσουμε να πετύχουν αυτούς τους δύο στόχους. Στη σημερινή κοινωνία πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη σημασία των φροντιστών σε κάθε οικογένεια. Το να φροντίζει κάποιον ε, σημαίνει μεγάλη δέσμευση και σωματική αλλά και ψυχική. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στους φροντιστές και να τους παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη. Πιστεύω επίσης ότι η πρόταση αυτή θα, όλα τα μέλη, θα ωφελήσει όλα τα μέλη της οικογένειας ε, που φροντίζει και, την, ε, ε, και τους συγγενείς αλλά και τους ηλικιωμένους. Και αυτοί έχουν δικαίωμα στη ζωή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα και γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει αυτά τα στοιχεία σε αυτό το νομοθέτημα και δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά και κυρίως τα γόρια θα μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των δύο γονιών. Αυτό θα βοηθήσει να αλλάξει η νοοτροπία και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να υποστηρίξετε αυτό το νομοθέτημα. Είναι ισορροπημένο, είναι καλό για τους άνδρες, για τις γυναίκες, για τις οικογένειες, αλλά και για την οικονομία. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Ευρώπη προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας. Και τώρα για την Επιτροπή Δικαιωμάτων Ανθρώπου και την Ισότητα των Φίλων η κυρία Κοσλόφ Καράγεβιτς. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά τη Επιτροπή Γυναικών ε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ολοκλήρωση αυτής της πολύ καλοδεχούμενης ε, προσπάθειας. Συγχαίρω τον κύριο Κάζα που ε, ήταν υπεύθυνο για το θέμα αυτό και ευχαριστώ και όλες τις οργανώσεις και φορείς που συμμετείχαν ε, πολύ επικοδομητικά στη διαμόρφωση της πρότασης αυτής. Η πρόταση αυτή επίσης συζητήθηκε στην Επιτροπή μας διότι το πρόβλημα ισότητας των φύλων δημιουργεί πολλέ δυσχέρειε για τις γυναίκες. Ε, οι γυναίκε κυρίω ασχολούνται με την οικογένεια. Οι γυναίκε παίρνουν άδεια όταν αρρωστούν τα παιδιά. Οι γυναίκες ε, διακόπτουν την εργασία του και πληρώνουν ένα πολύ ψηλό τίμημα. Και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανεί ότι οι γυναίκε ε, θυσιάζουν τη σταδιοδρομία του για τα παιδιά και αυτό έχει ω αποτέλεσμα η μέση σύνταξη των γυναικών να είναι 40% Χαμηλότερε από τι ε, συντάξει των ανδρών και οι, εργα... εργοδότες θεωρούν ότι οι γυναίκε ε, είναι λιγότερο διαθέσιμε ε, στον τόπο εργασία και γι' αυτό τείνουν να μην τι προσλαμβάνουν και αυτό είναι απαράδεκτο αυτή η νέα νομοθεσία θα ενθαρρύνει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση του χρόνου εργασία και θα οδηγήσει και σε καλύτερο επιμερισμό των καθηκόντων μεταξύ των γονέων παράλληλα θα ενισχύσει τη θέση των γυναικών αλλά έτσι και των ανδρών οι άνδρες θα έχουν το δικαίωμα να ανατρέφουν στο σπίτι τα παιδιά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό καθήκον. Αυτό φέρνει τα μέλη της οικογένειας πιο κοντά. Να μην ξεχνάμε τα πιο σημαντικά στοιχεία. Ελάχιστη διάρκεια γονικής άδειας δύο μήνες και επίσης η άδεια πατρότητας. Αυτή είναι μια πρόταση που είναι καλή για όλη την οικογένεια και γι' αυτό καλό όλες τις πολιτικές ομάδες να στηρίξουν αυτό το κείμενο να σταθούμε στο πλευρό των παιδιών, των γονέων και των οικογένειων. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. κύριε πρόεδρος. Και εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Τίσεν, η Επίτροπο έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί εισηγητέ, κυρίε και κύριοι, Καλωσορίζω την πρόταση. Χαιρετίζω τους κυρίους Κάζα και Κοσλόφσκα, συγητή και συνσηγήτρια, τους, τους και οδησηγητές και όλους όσοι αφοσιώθηκαν στην πρόταση αυτή οδηγία. Κάνατε ό,τι μπορούσατε για να βρείτε μια καλή συμφωνία. Μια καλή συμφωνία που δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την διάθεση συνεργασίας και τη βούληση συνεργασίας από πλευρά Κοινοβουλίου αλλά και Συμβουλίου και τη δική σας ε, αποφασιστικότητα να βρείτε μια λύση στις συνομιλίες. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και η δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο εξισορρόπησης του οικογενειακού με τον επαγγελματικό βίο ενισχύεται χάρη σε αυτήν την οδηγία. Ταυτόχρονα δίνεται και δυνατότητα στους πατέρες να μένουν με τα παιδιά τους. Γιατί αυτή τη στιγμή πατέρες και μητέρες αναγκάζονται να κάνουν επιλογές δύσκολες μεταξύ του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου και αυτό ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα βαρύ για τις γυναίκες. Οι στατιστικές στην αγορά εργασίας δείχνουν 11,5% ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη απασχολησιμότητα των γυναικών από ότι στον πληθυσμό των ανδρών. Αυτό σημαίνει επίσης 16% απόκληση με ε, αντανάκλαση στο συνταξιδοτικό κενό χάσμα η διαφορά σε ύψος 36%. Έτσι λοιπόν η πρόταση αυτή ε, λένε κάποιοι θα παρέμβει στον οικογενειακό προγραμματισμό ή τις προσωπικές επιλογές των οικογενειών. Όχι, εγώ θα πω ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η οδηγία στόχο έχει να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες, κίνητρα επιλογές στους συμπολίτε μας. Μόνοι τους θα αποφασίσουν ποια είναι η αγορά, ε, ποιος είναι ο συνδυασμός οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Οι γονείς οι ίδιοι θα μπορούν να κάνουν τις επιλογές αυτές. Έτσι, χάρη στην οδηγία θα υπάρχει συνολικά ε, τέσσερις μήνες γονεϊκή άδεια, εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον μήνες θα ανήκουν κατά τρόπο μη μεταβιβάσιμο και, κατάλληλο, και με κατάλληλο τρόπο στον ε, λόγο γονέα. Θα το οργανώσουν βέβαια αυτό τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι έτσι έχουμε βρει και μια καλή συμβαστική λύση από τον τριμερή διάλογο. Έχουν επιπλέον 10 ημέρε ε, πατρικής ε, άδεια οι πατεράδες και μάλιστα με αποζημίωση σε ύψος άδεια εργασία, άδεια ε, ασθενείας. Η οδηγία επίσης δίνει απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, στη γύρανση του πληθυσμού. Εισάγει δηλαδή άδεια για φροντιστή πέντε ημερών και αυτό επιτρέπει στους ε, συμπολίτες μας να φροντίσουν τους ε, οικείους τους. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, θεωρώ πως η οδηγία προσφέρει μια συγκεκριμένη, μια σαφή βελτίωση στη ζωή των συμπολιτών μας ε, μεταμορφώνει και υλοποιεί τις υποσχέσεις του κοινωνικού πυλώνα και μας προωθεί προς την υλοποίηση και των στόχων των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ για την προσήλωση και αποφασιστικότητά Σε Ευχαριστώ πολύ και τώρα οι ομιλητές εκ μέρους των ομάδων Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με την κυρία Μωρέα Σαρτιέ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα πρώτα μου λόγια είναι για την Επίτροπο, την κυρία Τίσεν. Θαυμάζω πάρα πολύ τα όσα κάνετε, κύριε Επίτροπε, μέσα από αυτό το κείμενο. Πρόκειται για ένα ε, πολύ μοντέρνο κείμενο και ήσασταν ε, θαραλέα ε, να βάλετε αυτό το κείμενο για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στο τραπέζι μας. Είναι ένα κείμενο που έρχεται να ανατρέψει τις πανάρχες συνήθειες που είναι εγγεγραμμένες στην κοινωνία μας όπου το άκθος, την ευθύνη της οικογένειας την έχουν μόνο οι γυναίκες και έρχεται ε, αυτό να μπλοκάρει τη σταδιοδρομία τους ε, και ακόμη και έχει τίμημα στην αγορά εργασίας. Και με αυτό το κείμενο έρχεστε να επανεξισορροπήσετε αυτή την αδικία που βιώνουν πάρα πολλές γυναίκες. Θα ήθελα να σας πω ευχαριστώ εξ ονόματος όλων αυτών των γυναικών. Και βέβαια ευχαριστώ και τον David Κάζα, τον εισηγητή μας, ο οποίος μπόρεσε να πάει μέχρι το τέρμα των πεποίθησεών του και ε, φυσικά ε, αυτή είναι η δουλειά του Ευρωβουλευτή, γιατί μπορεί να έχουμε ένα καλό κείμενο ε, επιτάπητος, μπορεί να έχουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ εισηγητή και σκιωδών εισηγητών, όμως αν δεν επικυρωθεί όλη αυτή η εργασία από αποτελεσματικού τριμερείς διαλόγους, δεν αξίζει τίποτα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς. Πρόκειται για ένα νέο λιθαράκι της κοινωνικής Ευρώπης που τίθεται στο τραπέζι μας σήμερα το πρωί και πρέπει να το επιστηρίξουμε. Πρόκειται για ένα νέο λιθαράκι που αλλάζει την αγορά εργασίας, που αλλάζει την έννοια της οικογένειας και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αγορά εργασίας αλλάζει γιατί Πράγματι βγαίνουμε από αυτό το ε, βάρος που πέφτει μόνο στη γυναίκα και θα έχουμε ισότητα ε, στους μισθούς και στη στιδιοδρομία. Και αυτό θέλουμε για τις γυναίκες. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ στους Δημοκράτες. Αρένα, δύο λεπτά και 30 δεύτερα. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με την ε, κυρία Μωρέν Σαρτιέ στις ευχαριστίες ε, απέναντι στην Επίτροπο αλλά και στον εισηγητή. Είναι αλήθεια ότι ζούμε ακόμη στον 21ο αιώνα, βιώνουμε εισαγωγή διακρίσεων, ιδιαίτερα διακρίσεις απέναντι στις γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές ε, που σήμερα δέχονται διάκριση στην απασχόληση, στη διαδρομία τους, αλλά και στους μισθούς. Οι λόγοι ο λόγος ε, θα έλεγα είναι απλώς επειδή μπορούμε να είμαστε μητέρες. Ο λόγος αυτής της διάκρισης είναι η ικανότητά μας ε, να γίνουμε μητέρες και να κοιοφορούμε. Θα έλεγα όχι μόνο το γεγονός ε, του να κάνουμε παιδιά, αλλά το να μπορούμε μία μέρα να έχουμε παιδιά. Αυτό αποτελεί παράγοντα διάκριση απέναντί μα και οι εργοδότε θεωρούν ότι είναι ένα κίνδυνο σε σχέση με την απασχόληση και τη σταδιοδρομία. Εννέα μήνε κοίηση θα δικαιολογούσαν σήμερα ένα χαμηλότερο ποσοστό απασχόληση από αυτό των ανδρών. Θα δικαιολογούσαν 16% διαφορά στου μισθού και θα δικαιολογούσαν 30% διαφορά στι συντάξει. Συνδυτοποιείται 9 μήνε στη ζωή ε, και μπαίνετε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό προτείναμε σήμερα μία λύση, μία από τις ε, ενδυνάμει λύσεις ε, που θα θέσουν σε ισότιμη βάση τους άντρες και τις γυναίκες. Είναι αλήθεια ότι μόνο με μία οδηγία δεν θα τα καταφέρνουμε. Δέκα μέρες για άδεια μετρότητας ε, δεν είναι ισότιμο με την άδεια μετρότητας, αλλά είναι κάτι. Το μεταβίβαστο της άδεια. Μιλήσαμε για το μεταβίβαστο στριμερείς διαλόγους για δύο μήνες. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Μπορούμε να πάμε πιο μακριά Κυρίω ό,τι αφορά του μισθού και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωση. Τώρα, πέντε μέρε για του φροντιστέ είναι μια νέα οδηγία. Ε, έτσι λοιπόν θέλω να πω ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τη δουλειά που κάνετε για αυτό το βήμα προ τον μπρο. Όμω ε, φυσικά θα πρέπει να ελέγξουμε την εφαρμογή αυτή τη οδηγία, γιατί ε, ουσιαστικά αποτελεί μια βάση και επομένω κάθε κράτο μέλο που αισθάνεται πιο γενναιόδωρο για περισσότερη ισότητα είναι ευπρόσδεκτο για την καταπολέμηση τη εισαγωγή διακρίσεων. Όμως έχουμε μια δουλειά να κάνουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε να επαγρυπνούμε ότι η οδηγία θα καταπολεμήσει όλες τις διακρίσεις που γίνονται σήμερα απέναντι στις γυναίκες στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ομάδα ICR, κυρία Ζητνότσκα. Ένα λεπτό και τριάντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά μιλάμε για την ισότητα ανδρών και γυναικών, συμμετοχή των γυναικών στον εργασιακό βίο, καλύτερη εξορρόπηση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Η πρόταση την οποία καλούμαστε τώρα να ψηφίσουμε ε, αποτελεί ένα καλό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων αυτών, προσδιορίζοντα ε, ελάχιστες προδιαγραφές Δηλαδή εισάγει ένα ελάχιστο επίπεδο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με παρκές επίπεδο ε, χειρισμών και διευθετήσεων για τα κράτη-μέλη ώστε να ορίσουν συστήματα που προσυδειάζουν στις εθνικές τους κοινωνίες. Εδώ εγώ πιστεύω προσωπικώς ότι πρέπει η μητέρα να μπορεί να μεριμνά για το νεογέννητο μωρό της αλλά και για κάποιον άρρωστο που ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία χρειάζεται φροντίδα. Αυτό διαφέρει όμως από αυτά τα οποία μπορέσαμε μέσα από τον τριμερή διάλογο να αποκομίσουμε. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε πιο πιο γενναιόδορη υποστήριξη. Αλλά, και είναι μεγάλο το αλλά, αυτή η επιλογή πρέπει να εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Πρέπει τα κράτη-μέλη δηλαδή να έχουν το, ε, την ελευθερία, τη διακριτική, ώστε να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Η πατρική άδεια επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούν οι πατέρες να ε, παίρνουν μερικές μέρες άδεια όταν γεννιέται το παιδί τους. Στη Σλοβακία το έχουμε συστήσει πολύ αυτό, αλλά δεν έχει γίνει τίποτε μέχρι τώρα. Μια άδεια για τους φροντιστές επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρόκειται για υποστήριξη πολύ σημαντική για τις οικογένειες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Για την άλλη, κυρία Βίβα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ο εισηγητής και οι σκιώδης ε, αξίζουν συγχαρητήριο για την εργασία τους. Αυτά που επιχειρήσαμε εναρμονίζονται με την φιλόδοξη προσέγγιση της Κομισιόν και την βελτιώσαμε ακόμη περισσότερο. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, το κείμενο όμω έχει αποδυναμωθεί. Θα ήθελα ισχυρότερα μέτρα για την άδεια πατρότητα στο επίπεδο ε, αμοιβών κατά την άδεια, τη γονική άδεια, γιατί οι μελέτες λένε σαφώς ότι περίπου το 85% των αμοιβών των εργαζομένων αποτελεί κίνητρο για να πάρουν και οι άνδρες ε, άδεια πατρότητας αλλά οι συνομοθέτες δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Πολλά λοιπόν ε, θα μείνουν στα χέρια των κρατών μελών. Και στο τέλος ε, η αλλαγή σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση είναι μικρή. Είναι ένα θετικό βήμα αλλά μικρό. Για την οδηγία των φροντιστών όμως ε, έχουμε πραγματικές καινοτομίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά τα κράτη-μέλη έδειξαν απροθυμία ή υπερβολική επιφυλακτικότητα. Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι η ευθύνη για την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ε, ασθενών ε, αναλαμβάνεται κυρίως από τις γυναίκες και αυτό έχει επιπτώσεις στην καριέρα τους, στην κοινωνική τους ζωή, τις αμοιβέ τους. Όμως το κείμενο και εδώ είναι ένα θετικό βήμα. Δεν πρόκειται για επανάσταση, αλλά τουλάχιστον ε, θα έχουμε αμοιβόμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο άδεια πιτρότητας, δύο μήνε γονική άδεια που δεν μπορεί να μεταφερθεί και πέντε μέρε άδεια για του φροντιστέ. Επιπλέον, οι πολίτε μα μπορούν να ζητήσουν ευελιξία στι συνθήκες εργασία, ούτω ώστε να μπορούν να συνδυάσουν καλύτερα την οικογενειακή με προσωπική ζωή και τι ε, ευθύνε του για τη φροντίδα. Ελπίζω να βελτιωθεί περαιτέρω στο μέλλον. Ευχαριστώ για την QNGL, κυρία Γκονθάλεθ Πένια. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι άδειε μητρότητα και πατρότητα πρέπει να έχουν την ίδια διάρκεια, να μην μπορούν να μεταφερθούν και να έχουν ε, αμοιβή 100% του μισθού. Αυτό θέλουμε και η προσωρινή συμφωνία απέχει πολύ από αυτό. Δεν μα ικανοποιεί. Εισηγάγαμε διάφορε τροπολογίε, πρώτα απ' όλα για να μην μπορεί να μεταφερθεί η άδεια αυτή. Αυτή είναι απαραίτητη προπόθεση για να υπάρχει ισότητα για τα άτομα που φροντίζουν ε, συγγενείς τους και για την αγορά εργασίας. Και η αμοιβή 100 ή 80% είναι απαραίτητη για να ε, μην σημαίνει φροντίδα ε, των παιδιών και των ηλικιωμένων και των ασθενών μείωση του εισοδήματο. Και δύο εβδομάδε γονικής άδεια πρέπει να είναι υποχρεωτικέ, γιατί πρέπει και οι δύο γονεί να ασχολούνται με τον νεογέννητο. Αυτό είναι κάτι το ελάχιστο βελτιώνει τη ζωή των ε, συμπολιτών μας. Ωστόσο, είχαμε δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα για να ε, βοηθήσουμε να υπάρχει μια κοινωνική Ευρώπη που να αγωνίζεται για την ισότητα. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω στην επόμενη θητεία να αναθεωρηθεί αυτό το κείμενο για να ε, βελτιωθεί ακόμη περαιτέρω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πράσινη τώρα. Ο κύριος Ουρτασούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κείμενο μα αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση. Είπαμε πολύ μακριά ε, από άδειε που δεν θα μεταφέρονται και θα πληρώνονται 100%. Όμω θα έχουμε ένα πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή πολλών πολιτών. Σε πέντε χώρε για πρώτη φορά θα έχουμε άδεια πατρότητα και σε οκτώ θα είναι μεγαλύτερη αυτή η διάδα από σήμερα και έχουμε βάλει και τέσσερι μήνε γονική άδεια και οι δύο δεν θα μπορούν να μεταφέρονται και θα πληρώνονται. Υπάρχουν μικρά βήματα λοιπόν προς τα μπρος ε, παρόλο που η ε, αμοιβή της, ε, πατρότητα, της άδειας πατρότητας είναι πολύ πιο κάτω από το 80% που θα ήταν το ελάχιστο που θα στείναμε και η γονική άδεια δεν έχει ελάχιστη αναφορά για την αμοιβή. Νομίζω λοιπόν ότι δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε και θέλω να ευχαριστήσω τον συγητή, του Σκιώδης και την Κομισιόν που ήταν πιο φιλόδοξοι σε σύγκριση με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο κάθε φορά που υιοθετούμε με ένα μέτρο του κοινωνικού πυλώνα δεν μπορούμε κάθε φορά να συζητάμε πόσο θα κοστίσει σε κάθε χώρα. Πρέπει να έχουμε φιλοδοξία για το μέλλον και θα ε, εργαστούμε στην επόμενη θητεία για να βελτιώσουμε αυτές τις διατάξεις. Ευχαριστώ. Η ευθυντή κυρία Μπεγκίν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όποια και είναι η ιδέα που έχετε σχηματίσει για το θεσμό τη οικογένεια, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα πράγμα πρέπει, μπορούμε να συμφωνήσουμε, πιστεύω. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι ούτε η μετανάστευση ούτε η τρομοκρατία, αλλά το να μπορεί να υπάρχουν οικογένειε και στο μέλλον, δηλαδή να συνεχίσει να υπάρχει η Ευρώπη. Οι τελευταίε δημογραφικέ ε, έρευνε δείχνουν ότι θα καταρρεύσει ο, δημογραφικά ο ευρωπαϊκό πληθυσμό μέχρι το 2050 και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε αυτή την τάση. Έτσι λοιπόν, εάν δεν εγγυηθούμε ε, δικαιώματα στους εργαζόμενου και προστασία για τους νέους δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Πρέπει να προσφέρουμε λοιπόν στους νέους και τις γυναίκες τη δυνατότητα να έχουν καλύτερες ε, συνθήκες εργασίας και να συνδυάσουν καλύτερα τον επαγγελματικό με τον οικονομικό βίο. Η οδηγία λοιπόν και με την άδεια την πατρική που προτείνει για τις ε, ε, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μέχρι 10 ημέρες τουλάχιστον ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχει επίσης η γονική άδεια μη μεταφέρσιμη με δύο μήνες με πλήρη μισθό που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνονται μόνο οι μητέρες με τη μερίμνα για τα παιδιά. Επιπλέον έχουμε ζητήσει και έχουμε εξασφαλίσει πιο ευέλικτα ωράρια με την δυνατότητα της χρήσης και της τηλεαπασχόλησης έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των οικογενειών και κυρίως τη φροντίδα για τους αναπήρους ή ε, αρρώστους ε, οι εργαζόμενοι. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πιο αυτόνομες ε, δομέ δομές προστασίας, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, για την παροχή φροντίδας στο σπίτι, εξειδικευμένης φροντίδας, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να συνδυάζει και την επαγγελματική του σταδιοδρομία, αλλά και την ε, προσφορά υπηρεσίας και φροντίδας στα μικρά παιδιά ή τους ηλικιωμένους ή ασθενείς συγγενείς. Χωρίς να έχουμε επιτύχει όλα αυτά τα οποία επιδιώκαμε, βλέπουμε ότι μπορούμε να, κάνουμε, να αποτιμήσουμε θετικά αυτή την πρόταση οδηγίας, γιατί βοηθάει και στην εξασφάλιση ε, συγκερασμού επαγγελματικού και του βίου και στην ανατροπή τη ε, πορεία προ την κατάρρευση που έχει πάρει το δημογραφικό στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι γνώμη και αν έχετε για το θεσμό τη οικογένεια, υπερψηφίστε τη για να συμβάλλετε έστω και λίγο σε αυτή την πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Μελά η ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτός ο φάκελος ε, για ε, του εργαζομένου και αφού αφορούν την ιδιωτική ζωή δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο πραγματικό τη στόχο δηλαδή να μπλέκεται σε κάθε στιγμή τη καθημερινή ζωή, των εργαζομένων στη γέννηση των παιδιών, την εκπαίδευσή τους ε, και στην βοήθεια που προσφέρει στους γονείς οι Βρυξέλλες ε, σε αντίθεση, μεταξύ, σε αντίθεση με αυτό που ανακοινώνεται για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή προκαλεί ανισορροπία γιατί πίσω από αυτή την ιδέα υπάρχουν υπάρχουν τρεις κίνδυνοι. Όλα τα νομοθετικά διοικητικά κείμενα στον τομέα αυτό ε, δεν ε, είναι παραρμοδιότητα των κρατομελών. Οι Βρυξέλλες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να θέτουν ε, ποσά, ποσοστά ή διάρκεια γιατί αυτό άπτεται τη αρχή τη επικουρικότητας και έρχεται σε αντίθεση με την ε, νομοθεσία της Γαλλίας όπου έχουμε όλη την απαραίτητη νομοθεσία. Επίσης αυτές ε, οι διατάξεις ε, δεν ικανοποιούν τους εργοδότες στο ρόλο να παρέχουν επαγγελματικές δραστηριότητες σε ένα αποδεκτό περιβάλλον και να μην επιβάλλουν υποχρεωτικό πατερναλισμό. Όμω, από ό,τι φαίνεται το κείμενο αυτό επιβάλλει την υπεροχή της ιδιωτικής ζωής ένα απέναντι της επαγγελματικής και ε, αυτό θα πλήξει την οικονομική δυναμική της Ευρώπης και καταρχήν θα πλήξει τις μισές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μη εγγεγραμμένος τώρα ο κύριος Φουντούλης το λόγο για ένα λεπτό. Η δημιουργία οικογένεια αποτελεί τη σημαντικότερη ίσω στιγμή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Επιπλέον είναι ο τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η συνέχεια των εθνών μα ω εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύεται με κάθε τρόπο και να ενθαρρύνονται οι νέοι να αποφασίσουν να κάνουν το μεγάλο αυτό βήμα. αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για όσου εργάζονται. δεν μπορούμε άλλο να επιτρέψουμε να τιμωρείται εργασιακά η δημιουργία οικογένεια ούτε να αναλαμβάνει περισσότερα βάρη ο ένα από του δύο γονεί είτε ο πατέρα είτε η μητέρα. συμφωνούμε απόλυτα λοιπόν με τη θέσπιση πανευρωπαϊκά του δικαιώματο γονική άδεια και για του δύο γονεί. επιπλέον θεωρούμε πω πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε και νομοθετημένε δυνατότητε ελαστικού ωραρίου και αδειών για του γονεί μέχρι την ηλικία εκείνη τα παιδιά θα μπορούν να εξυπηρετούν μόνα τους σημαντικό μέρος των καθημερινών τους αναγκών και συγκεκριμένα για εμάς μέχρι τα 12 έτη. Τέλος, ιδιαίτερη μέρημνα πρέπει να δοθεί στους γονείς παιδιών με ειδικέ ανάγκες, καθώς αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις σε σχέση με τους υπολείπους, καθώς και άδεια φροντίδας για εργαζόμενους φροντίζουν συγγενή που πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Ευχαριστώ. Και τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές. Πρώτα απ' όλα δύο λεπτά για την κυρία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αν εμεί ε, θέλουμε μια πιο κοινωνική Ευρώπη, αυτή η Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσει στι νέε απαιτήσει τη νέα κοινωνία. Και η κοινωνία αυτή είναι μια κοινωνία όπου οι οικογένειε ε, κάνουν όλο και πιο αργά παιδιά και οι γυναίκες είναι όλο και πιο ενεργές ε, στον εργασιακό κόσμο και οι άνδρες, οι πατεράδες επίσης ε, απαιτούν ε, να έχουν δικαίωμα στην πατρότητα και πολύ καλά. Εμείς βλέπουμε ότι στην Ευρώπη είχαμε πολύ μεγάλη απόκληση μεταξύ των δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν καλύπτουν τις οικογενειακές ανάγκες. Ε, τα ζευγάρια δυσκολεύονται να ανατρέψουν ε, τα παιδιά τους, όχι μόνο ε, όταν γεννιούνται, αλλά και στη σχολική ηλικία. Οι ανάγκες των παιδιών δεν συνάδουν με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό έχει οδηγήσει στην γύραση του πληθυσμού και στη μείωση της γεννητικότητας. Από την άλλη, αυτή η γενιά που έχει παιδιά όλο ένα και αργότερα είναι μια γενιά σάντουιτ, γιατί όχι μόνο πρέπει να προσέχει τα παιδιά, αλλά πρέπει να φροντίσει και τους γονείς της. Η γύρανση ε, στην Ευρώπη φέρνει αυξημένες ευθύνη ε, και θα πρέπει να ε, προσφέρουμε στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να μείνουν στο σπίτι με ε, μεγαλύτερη στοργή και τα ε, παιδιά τους δεν έχουν το δικαίωμα να μπορέσουν ε, να φροντίσουν όπως πρέπει τους γονείς τους. Γι' αυτό επιγόντως θα πρέπει να δώσουμε μία εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν πήγαμε τόσο μακριά όσο οι προτάσεις που είχα παρουσιάσει, όμως είμαι βέβαιη ότι αυτή είναι μία πρόκληση της κοινωνικής Ευρώπης για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπλίνκε Βιτσιούτε. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα Εγκρίνοντας αυτή την οδηγία νομίζω ότι στέλνουμε ένα καλό μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά ή ε, όσους φροντίζουν ηλικιωμένους ή ασθενείς. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι γυράσκει η Ευρώπη και πρέπει να δώσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για να επιτρέψουμε στους εργαζόμενους ε, να φροντίσουν για όλα τα άτομα και έτσι θα αυξήσουμε και τη γεννητικότητά μας πιστεύω. Είναι σημαντικό και οι γονείς ε, να έχουν άδεια πατρότητας. Αυτό θα βελτιώσει την ισότητα ευκαιριών για τις γυναίκες να έχουν περισσότερες δυνατότητες ε, στην σταδιοδρομία τους. Βεβαίως οι δικέ μα προθέσει ε, ήταν πολύ πιο φιλόδοξε από τη στάση των κρατών μελών, αλλά καλωσορίζω τη συμφωνία που επετεύχθη μετά από τι διαπραγματεύσει. Έτσι, κάθε πατέρα θα μπορεί να έχει 10 μέρε άδεια όταν γεννιέται το παιδί του. Θα έχει λοιπόν ε, και τη δυνατότητα να μοιραστεί την γονική άδεια με τη μητέρα για να αναθρέψουν και οι δύο να φροντίσουν τα παιδιά τους. Και έχουμε και για πρώτη φορά μια ευρωπαϊκή άδεια πέντε μερών για τα άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους ή ασθενείς συγγενείς τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι το εργασιακό περιβάλλον φιλικό προς τις ανάγκες της οικογένειας όλες αυτές, ούτως ώστε οι εργοδότες να διασφαλίζουν ευέλικτες συνθήκες εργασίας και αυτό πιστεύω ότι θα βελτιώσει ε, και την υγεία των μελών της οικογένειας. Ευχαριστώ την Επιτροπή για το πόσο έβαλε σε αυτήν την εργασία. Ευχαριστώ ο κύριος Χοκ. Ε, ε, ο Κομφούκιος είπε να επιλέξεις μια εργασία που αγαπάς και δεν θα εργαστείς ποτέ στη ζωή σου. Ένα άτομο που είναι ικανοποιημένο στην ε, ιδιωτική του ζωή θα είναι πολύ πιο χαρούμενο και στον χώρο εργασίας του. Πρέπει λοιπόν να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο πλευρών της ζωής ενός ανθρώπου. Αλλά η οδηγία αυτή έχει βέβαια κάθε λόγο να υπάρχει, είναι πολύ θετική, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση στην οικογενειακή ζωή. Με βάση το Πολωνικό Σύνταγμα, όλη αυτή οι τομεί όμω είναι η ειδική φροντίδα του κράτου. Παρ' όλα αυτά, να μην ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να θεωρούν ότι παρεμβαίνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβολικά σε οικογενειακά θέματα και το οικογενειακό δίκαιο. Ορισμένες από τις διατάξεις είναι βεβαίω συμβατέ με την δική μας νομοθεσία. Αλλά, για παράδειγμα, στην Πολωνία εμείς προβλέπουμε 14 μέρες ε, άδεια πατρότητας κατά τη γέννηση τέκνου. Οπότε με αυτό συμφωνούμε. Αλλά δεν θεωρούμε ότι χρειάζονται αναγκαία δύο μήνε και ότι πρέπει να υπάρχει μη φορητότητα. Ευχαριστώ κύριο Καλβέτ Τσαμπόν. Ένα... Ευχαριστώ, Λόεδρα. Κύριε Επίτροπε, καλημέρα. Θα ήθελα να συγχαρώ όλου του κοιόδη εισηγητέ και φυσικά τον κύριο Κάσα, τον εισηγητή, που έχουν εκπονήσει ένα πολύ σημαντικό κείμενο για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τους εργαζομένους. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλού εργαζομένου. Όμω, προφανώ, αυτό το κείμενο αποτελεί ένα βήμα και όχι μικρό, ένα σημαντικό βήμα που προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, που ε, μειώνει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ε, και ε, προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή. Θέλω να επιμείνω στο πώς αυτό ε, γράφεται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα και είμαι πολύ ικανοποιημένος ε, και συγχαίρω και την Επίτροπο ε, που συμμετέχουμε σε αυτή την οδηγία που παρέχουν βασικά δικαιώματα για την κοινωνική συνοχή. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Ουρτασούν πριν. Σίγουρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να ε, σημειώνουν πρόοδο σε αυτό, όμως η πρόκληση για την επόμενη θητεία είναι να έχουμε μία αλληλεγγύη τη Ευρώπη για το κοινωνικό. Καλημέρα σας, η κυρία Κούνεβα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Γονιός, πώς να ορίζετε άραγε είναι το τόξο από το οποίο τα παιδιά σαν ζωντανά βέλη ξεκινάνε να πάνε μπροστά. Έγραψε στο ποίημά του προφήτης ο Χαλίλ Γκυμπράν. Η οδηγία για την εξισορρόπηση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής δεν είναι αυτή που φανταζόμουν όταν ξεκίνησα να δουλεύω αυτόν τον φάκελο. Δυστυχώς δεν αναθεώρησε την άδεια μητρότητας παρά τις πιέσεις μας. Ρυθμίζε δε ελάχιστα τις άδειε για τους γονείς που εργάζονται. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα που θα επιτρέψει σε εκατομμύρια γονείς στην Ευρώπη να είναι στη ζωή των παιδιών τους σήμερα ώστε να είναι στις αναμνήσεις τους αύριο για αυτό το αύριο δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε για μια Ευρώπη κοινωνικότερη, δικαιότερη, για μια Ευρώπη το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση για την, τον συνδυασμό επαγγελματικού και κοινωνικού βίου ήταν ε, ε, αναμενόμενη για καιρό και όχι μόνο γιατί περιμέναμε να βγει αυτή η συμφωνία με την ένταση της διαδικασίας των συνομιλιών, μιας διαδικασίας που ναι, κράτησε κάποια χρόνια. Ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω ότι βελτιώνονται χάρη στις τελευταίες ε, ρυθμίσεις ε, τα στοιχεία του πλαισίου, χωρίς ωστόσο να έχουν φτάσει στο αρχικά τόσο φιλόδοξο ε, επίπεδο της εντολής που είχαμε για τη διαπραγμάτευση. Θα θέλαμε κάτι πολύ καλύτερο βεβαίως, αλλά ως πολίτης και πατέρας μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος έστω που έχουμε την εισαγωγή της πατρικής άδεια σε ευρωπαϊκό κείμενο με 10 ημέρες. Ε, διάρκεια, όχι όμως, ε, κρίνω όμως όχι επαρκή την αποζημίωση σε όρους ε, άδειας ασθενείας. Η γονεακή άδεια είναι μια από τις, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε, στην τρέχουσα θητεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Τσόκα, ένα λεπτό και τριάντα δεύτερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά κάνει και προχωρεί προ μια στρατηγική κατεύθυνση για το συνδυασμό του επαγγελματικού και του, οικονομικού, του οικογενειακού βίου. Μια κατεύθυνση σωστή βεβαίως Πρέπει να επενδύσουμε στις αξίες της οικογένειας, στην αξία της οικογένειας αλλά και στην ανάπτυξη εκ νέου της γενετικότητας για την κοινωνία και την Ευρώπη και για τη χώρα την ίδια. Ο συνδυασμός οικογενειακού και επαγγελματικού βίου βοηθά τους ε, άνδρες της γυναίκες, στην οικονομία της Ιταλίας, στην οικονομία της Ευρώπης συνολικά για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό κενό τα κενά λίκνα όπως λέμε. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε εμπιστοσύνη στο συνδυασμό σε αυτές τις ε, περιοχές οι οποίες έχουν ε, κατά τρόπο υποδειγματικό όπως η Λομβαρδία παραδείγματι ε, και πρωτοποριακό εισαγάγει μέτρα που δίνουν συγκεκριμένα λύσεις συνδυασμού του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Η περιφέρεια της Λομβαρδίας έχει τα τελευταία χρόνια επενδύσει 30 εκατομμύρια και για βρεφονιπιακούς σταθμούς και για άλλες μονάδες μέρημνας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε στις αρχές τις αρμόδιες στο πιο εγγύστο πολίτη επίπεδο να δώσουν τις απαντήσεις όπως έπραξε και η περιφέρεια της Λομβαρδίας. Αποτελεσματικές λύσεις για το συνδυασμό του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Ευχαριστώ κυρία Σόιντροβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κυρία Επίτροπε, Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ ευχάριστο για σας ε, να ακούτε τόσους επένους ε, για αυτή την ε, οδηγία και επίσης επένους για τους τριμερείς διαλόγους. Σίγουρα κάποιοι ήταν πιο φιλόδοξοι, κάποιοι ήταν κατά, αλλά τελικά βρήκαμε ένα συμβιβασμό που φαίνεται ότι είναι καλός για όλους είναι κάτι που θα υποστηρίξει τους γονείς και τις οικογένειες. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση αυτή και θέλω να τονίσω τέσσερα σημεία που είναι σημαντικά για μένα για να υποστηρίξω αυτή την οδηγία. Κατερχήν, ε, ελάχιστο δύο εβδομάδες ε, Άδεια πατρότητα, δύο μήνε, γονική άδεια, μη μεταβιβάσιμη, ευέλικτε ρυθμίσει εργασία και η άδεια των φροντιστών. Αυτά είναι τα ελάχιστα πρότυπα επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε. 28 κράτη-μέλη με διαφορετικέ παραδόσει και διαφορετικά συστήματα. Αυτά είναι λοιπόν τα ελάχιστα στα οποία μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή η οδηγία είναι ένα ισχυρό μήνυμα προ τα κράτη-μέλη ότι τα παιδιά αποτελούν επένδυση για το μέλλον. Τα παιδιά είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους γονείς στην υλοποίηση των ευθυνών τους. Εύχομαι στο μέλλον να έχουμε περισσότερο κατά νου τη δουλειά των γονέων. Αν μένει στο σπίτι με το παιδί σου και αυτό δουλειά είναι και θα πρέπει να σεβαστούμε και αυτή τη δουλειά. Πρόκειται για ένα καθήκον για τα κράτη-μέλη. Όλοι οι γονείς θα έπρεπε να έχουν μια ελεύθερη επιλογή και θα έπρεπε να αισθάνονται ότι η κοινωνία του σέβεται, αλλά και το κράτος. Αυτό αποτελεί επένδυση για το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ανυπομονώ για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας για να βοηθήσουμε τις οικογένειες και τα παιδιά. Γιονγκέριος, ένα λεπτό, Έχεις λόγο. ως γονιός Φυσικά θέλεις να κάνεις ό,τι μπορείς για να ξεκινήσει τη ζωή του με τον καλύτερο τρόπο το παιδί σου. Ως κόμμα PVDA θέλουμε όλοι οι γονείς να έχουν δυνατότητα να δώσουν στα παιδιά τους την αγάπη τους όταν γεννιούνται και να μην έχει να κάνει με το πόσα λεφτά έχεις ε, ή σε ποια χώρα ζεις. Δυστυχώς οι χαμηλόμιστοι γονείς δεν μπορούν να πάρουν αυτή την άδεια γιατί θα σημαίνει ότι θα μειωθεί πολύ το εισόδημά τους. Ε, γι' αυτό χαιρόμεθα που επιτύχαμε μια καλή συμφωνία και τώρα οι υπουργοί μας θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το κείμενο γιατί οι σωστοί κανόνες για την άδεια καθορίζουν ότι οι μητέρες θα πρέπει να κάνουν πολλά, θα πρέπει να μπορούν να βοηθούν και οι πατέρες και οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουν μαζί το παιδί τους όταν γεννιέται. Αυτό δημιουργεί ένα δεσμό μεταξύ γονών και παιδιών και ένα καλύτερο, μια καλύτερη μοιρασιά των καθηκόντων και επιτρέπει και στις γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Είναι ένα βήμα προς την κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και τώρα βίστησαν παρακαλώ Ισία. Πρόεδρε. Έχουμε με την νομοθεσία αυτή φτάσει σε νέα βάθη της παρέμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης με υποκρισία πάνω απ' όλα γιατί προσπαθείτε να υπαγορεύσετε σε άνδρες και γυναίκες πολίτες πώς πρέπει να, να φέρονται οι οικογένειες, πώς πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά τους. Εμεί θεωρούμε ότι οι αρμοδιότητες για τα θέματα της κοινωνίας ορίζονται από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη που εισπράττουν το φόρο έχουν και την ευθύνη για τα επιδόματα. Έτσι, απερίφραστα απορρίπτουμε την ανάμειξη της Ευρώπης σε θέματα της κοινωνίας, σε θέματα που επηρεάζουν τη ζωή της οικογένειας, περιορίζοντας έτσι και το περιθώριο επιλογών των κρατών μελών και της κράτους προνοίας. Ο Πιμέντα. Η πρόταση αυτή οδηγία αποτελεί ένα παράδειγμα κοινωνική υπαναχώρηση ε, και εκμετάλλευση με υποχρεωτική περίοδο άδεια. Ο ορισμό ε, τη αμοιβή βάση του επιδόματο ασθενεία ε, και η αποδοχή που γίνεται σε σχέση με τους φροντιστές. Είναι κάτι αρνητικό. Εδώ ε, ουσιαστικά σεβόμαστε τις ανάγκες των εργοδοτών ε, και δημιουργεί μια τυπολογία αδειών με μορφή που μπορεί να ε, αποτρέψει το χάρη προσωρινούς εργαζομένους από το να ζητήσουν άδεια. Η οδηγία αυτή δεν επερασπίζει τους γονείς αλλά τους εργοδότες οι οποίοι θα καθορίζουν πότε μπορούν να υποφεληθούν από τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι. Εμείς θέλουμε τη διεύρεση της άδειας να υπάρχει 100% αμοιβή, να ε, υπάρχει προώθηση πολιτικών υπέρ της μητρότητας, κάτι που απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς έτσι θα καταψηφίσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ. Ράιντ και για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τώρα που ξεκινάει η προεκλογική εκστρατεία λέγονται πολλά ψέματα για τις οικογένειες στην Ευρώπη. Ψέματα ότι δηλαδή για να προστατεύσουμε τις οικογένειες πρέπει να κάνουμε κηρύγματα μίσους κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ, να περιορίσουμε τα γεννόματα των γυναικών και να επιβάλλουμε μια ενιαία αντίληψη για το τι σημαίνει οικογένεια. Στη Βερόνα έγινε σαφές ότι υπάρχει μια συμφωνία ακραίων χριστιανών, συντηρητικών και ακροδεξιών που θέλουν να διαδίδουν τέτοια ψέματα. Το αντίθετο ισχύει. Για να προστατεύσουμε τις οικογένειες δεν χρειάζεται να είμαστε ομοφοβικοί και κατά των τρανς. Πρέπει να ε, στηρίξουμε τις οικογένειες. Όλες οι οικογένειες πρέπει να έχουν χώρο και αυτές για την κοινωνία. Πρέπει να αγκαλιάσουμε κάθε μορφή οικογένειας και θα πρέπει να υπάρχει χρόνος για να φροντίζουν τα μέτρα της οικογένειας τα μεν δε. Αυτή η οδηγία είναι σημαντικό κείμενο και είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σάντερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ο χρόνος ε, είναι αγαθό, πολύτιμο, έναν ανεπαρκία αν είναι κανείς γονιός ή φροντίζει άλλους. Έξι στους δέκα γονείς δεν μπορούν να επιτυγχάνουν αυτό τον, ε, την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και οικογενειακής της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και ε, αντιμετωπίζουν πολλές φορές κίνδυνο υπερκόπωσης και γι' αυτό η Ευρώπη θα, θα πρέπει να παίξει το σωστό ρόλο εκφράζοντας σωστά την ε, αλληλεγγύη προς την οικογένεια. Αυτοί είναι οι κανόνες που υιοθετούμε σήμερα. Είναι η απάντηση μιας Ευρώπης που δράσει συγκεκριμένα. Παρά τις διαφορές μας, χαίρομαι ιδιαίτερα που καταφέραμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί και να υπάρξει αυτό το ελάχιστο επίπεδο κοινωνικών κανόνων που θα συμβάλλει στην καλύτερη ζωή των οικογενειών, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κοινωνίας, Εισάγουμε λοιπόν ευρωπαϊκή άδεια πατρότητα για να εγγυηθούμε ότι όλοι οι πατέρε θα είναι παρόντε όταν γεννιούνται τα παιδιά του. Επίση, έχουμε και αυτή τη μη μεταφερσιμότητα για ένα τμήμα τη γονική άδεια. Ένα άλλο στοιχείο αυτών των νέων κανόνων είναι η εισαγωγή αυτή της άδεια για αυτούς που φροντίζουν συγγενείς. Γιατί έχουμε πολλούς ηλικιωμένους, πάνω από 20% των Ευρωπαίων είναι άνω των 65 επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες για λόγους επιλογής ή επειδή κοστίζουν πολύ αυτές οι υπηρεσίες, το 85% των φροντίδων για τα άτομα που έχουν ανάγκη είναι από συγγενείς τους. Να έχουν δυνατότητα κάποια άδεια είναι μια σωστή αμοιβή για την προσπάθεια που κάνουν που είναι τόσο αξιόλογη. Έτσι κάνουμε ένα πρώτο αλλά ουσιώδες βήμα και τώρα εναπόκειται στα κράτη-μέλη να κάνουν και αυτά, αυτά που πρέπει, δημιουργώντας για παράδειγμα χώρους που μπορούν να αναπαύονται τα άτομα αυτά, που φροντίζουν άλλα, για να μπορέσουν να ξαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιλσκογ, Μαρίτα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούστηκε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι κάποιες νομοθεσίες μπορούν να είναι περίτες. Το 1992 είχαμε μια πρώτη οδηγία όταν ήταν οι οικογενειακές δομές διαφορετικές στις διάφορες χώρες και αντίστοιχες νομοθεσίες ε, όχι αρκετά ανεπτυγμένες. Αυτό που κάνουμε εδώ όμως σήμερα έχει να κάνει με μια θεμελιώδη επιλογή που θα επιτρέψει ε, την ομαλή λειτουργία των οικογενειών και των κοινωνιών μας. Έχουν το δικαίωμα οι πατεράδες να βρίσκονται στο σπίτι, να συμβάλλουν στην ε, ανατροφή των παιδιών τους είναι λίγες οι γυναίκε που έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ε, κατά τρόπο ικανοποιητικό στην Ευρώπη, ενώ χρειαζόμαστε όλο αυτό το εργατικό δυναμικό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε περισσότερη ισότητα στην κοινωνία που είναι ουσιώδη και για την οικογένεια, το άτομο, το παιδί, την οικονομία. Και γι' αυτό μιλούμε σήμερα. Αυτό είναι το εγχείρημά μα. Η κυρία Στέβεν, σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία κατάλληλη ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή ε, είναι ζωτική. Όλοι εμεί, ε, ιδίω οι γυναίκε, θα πρέπει να έχουμε ευκαιρίε ε, στην αγορά εργασία. Οι γυναίκε συχνά πρέπει να διαλέξουν μεταξύ στεδιοδρομίας και ανατροφής των παιδιών, οικογενειακών καθηκόντων. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουν τις ανάγκες των πολιτών τους στην Φλάνδρα. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, καλή νομοθεσία ε, για την άδεια των φροντιστών η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει να επιβάλλει πράγματα στις εθνικές αρχές μπορεί να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Θα πρέπει να δει κανείς και τη θέση των εργοδοτών οι οποίοι ε, ουσιαστικά επιβαρύνονται η κυρία Ματέρα για ένα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Κάσα και την Αγνιέσια Κοσλόσκα για τη δεσμευσή τους και επειδή εργάστηκαν σε ένα κείμενο που επιτέλους θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Είναι σημαντικό κυρίως για τις ε, γυναίκες ε, ε, οι οποίες απλώς επειδή γίνονται μητέρες ή επειδή πρέπει να φροντίσουν συγγενείς δεν μπορούν να συμμετέχουν στον εργατικό βίο. Βάσει του εξυγχρονισμού ε, του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία θέλει να δώσει στους γονείς και στους φροντιστές τη δυνατότητα να συμφιλιώσουν την επαγγελματική και ιδιωτική τους ε, ζωή. Βασίζεται σε εφιστάμενα δικαιώματα η οδηγία και τα ενισχύει, εισάγοντα και διατηρώντα το επίπεδο προστασίας που, παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όμως ε, η έλλειψη άδεια πατρότητας με παροχές σε πολλά κράτη-μέλη οδηγεί ε, στο να μην χρησιμοποιούνται οι άδειε αυτέ από του ε, πατεράδε. Ευχαριστώ λοιπόν του συναδέλφου για τη δέσμευσή του να ανατραπεί η τάση αυτή. Υποστηρίζω λοιπόν ε, την ισορροπημένη προσέγγιση όταν δεν θίγονται τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Παροτρύνω του συναδέλφους εδώ να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή γιατί βελτιώνει την ισότητα των δύο φύλων εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί υποστήριξη των γυναικών στην επανάταξή του στην αγορά εργασία. Κάντε το για όλους τι μητέρε, του πατέρε και για τι μελλοντικέ γενιέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζεντήλε, παρακαλώ Ελένα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε το παράδειγμα του διαχωρισμού των ρόλων ε, είναι ε, περιορισμένο και ε, ουσιαστικά επιβάλλεται στις γυναίκες να συνεισφέρουν στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Αυτή είναι η στιγμή της ανάληψης ευθυνών του επιμερισμού των ευθυνών του χρόνου, της κούρασης, της χαράς, της φροντίδας και της οικογενειακής στοργής Καθώ ε, Καθώς η οικογένεια αποτελεί κοινότητα. Από τις σελίδες αυτής της οδηγίας αναδύεται η νέα Ευρώπη. Διαφαίνεται πολιτική και πολιτισμική αλλαγή για να ευνοηθούν ε, οι γονείς και γιατί ζητείται μια νέα ευθύνη από τους θεσμούς και τις επιχειρήσεις προκειμένου η συμφιλίωση να γίνει μια ευκαιρία ε, μέσω από τα οργανωτικά μοντέλα και διαφυλάσσοντας τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Βυσνιεύσκα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, η ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά. Και γι' αυτό πρέπει να βρούμε λύσεις που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε καλύτερα αυτήν την ισορροπία. Αλλά Ποια είναι αυτή τη στιγμή η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του προσωπικού μας εδώ, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το προσωπικό μας πρέπει να, έρθουν, πρέπει να έρθει στις 9 το πρωί το αργότερο και φεύγουν από το κτίριο αργά το απόγευμα. Τα δικά τους τα παιδιά ποιος τα φροντίζει. Τα ανατρέφουν οι παιδικοί σταθμοί και άλλοι τέτοιοι θεσμοί. Όταν ήταν έγκυος η βοηθός μου, εγώ είδα πώς θα μπορούσε να έχει ευέλικτες συνθήκες εργασίας και ε, αν θα μπορούσε να εργαστεί από το σπίτι και δεν το εφαρμόζουμε αυτά τα οποία προτείνουμε. Ε, ο κύριος Ντέτχεν, η Ευρώπη μπορεί να είναι κοινωνική μόνο αν υπάρχει ισότητα ευκαιριών και στο σπίτι και στο χώρο εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ομάδα μου καλεί εδώ και καιρό για περισσότερη ισορροπία, για τη φροντίδα και για την ανατροφή των παιδιών. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός ε, Πυλώνας το προβλέπει. Με την οδηγία που συζητάμε σήμερα επιδιώκουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Έτσι θα συμβάλλει η Ευρώπη για μια σύγχρονη φροντίδα και ανατροφή και θα πρέπει να γίνει καλύτερη κατανομή των καθηκόντων εντό τη οικογένεια. Τουλάχιστον τέσσερι μήνε γονική και δύο από αυτού δεν θα, μπορούν να, δεν θα πρέπει να μπορούν να μεταφερθούν. Αυτό θα είναι επαρκές κίνητρο να αναθρέφουν και οι πατέρες τα παιδιά τους. Αυτό το λέμε πολύ συγκεκριμένα. Με αυτή τη νέα προσέγγιση και οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 10 μέρες άδεια πατρότητας και οι 5 μέρες άδεια για τους φροντιστές αμοιβόμενες είναι πολύ θετικό όμως δεν επαρκούν όλα αυτά στην Ιρλανδία το ποσοστό είναι μόνο 36% για παράδειγμα της αμοιβή που θα λαμβάνουν σε σχέση με την κανονική αμοιβή του. Δεν είναι επαρκές αυτό που επέβαλε λοιπόν το Συμβούλιο και αυτό δεν με ικανοποιεί και ευχαριστώ πολύ. Σάιμον, παρακαλώ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το μέτρο αυτό προτάθηκε πριν από δύο χρόνια. Πέρασε πέντε μήνες σε τριμερή διάλογο. Είναι ξεκάθαρα από αυτού του τύπου τα νομοθετήματα που δεν δίνουν μία λύση ομοιόμορφη για όλου, αλλά προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία στα κράτη-μέλη να διατυπώσουν το καθένα τη δική του νομοθεσία με βάση τα δεδομένα, τι παραδόσει του, αλλά και ταυτόχρονα η ήπια ανεβάζει τον πύχη για τους πάντες. Έτσι λοιπόν και τα πιο πλούσια ε, κράτη ή τα κράτη που έχουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξασφαλίσουν περισσότερη προστασία για τους πολίτες τους χωρίς να τους υποδεικνύουν οι εντό αγωγικών ευρωκράτες το τι θα κάνουν. Έτσι λοιπόν και οι γονείς και οι φροντιστές θα έχουν μεταποδοχών άδεια εάν μείνει βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο και στη διαδικασία Eye τώρα η κυρία Κινίτσι Κατερίνα. Σε παρακαλώ να λάβεις το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η οδηγία που συζητούμε σήμερα συμβάλλει θετικά στην κάλυψη των ε, ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, συνδυάζοντας καλύτερα τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό βίο για άνδρες αλλά και γυναίκες έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν και εκείνες ε, την σταδιοδρομία τους όπως το επιθυμούν πλήρως. Έτσι, προδιαγραφές ε, ορίζονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ελάχιστες βέβαια για την γονεακή αλλά και την πατρική άδεια, με ελάχιστο επίπεδο ε, αμοιβή και τις άδειες που ε, μπορούν να παίρνουν οι πατέρες ώστε τα παιδιά να μην είναι αποκλειστική φροντίδα των ε, μητέρων. Βεβαίως ε, θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τις δυνατότητες εκείνες της απασχόλησης τους γονείς αλλά και την πρόσβαση στις υποδομές υποδοχής παιδιών και φροντίδας για εξαρτημένα άτομα που θα επιτρέψουν στις οικογένειες να συνδυάσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό βίο. Είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν την υπηρεσία τους φροντιστές στους οικείους τους. Ευχαριστώ Σολέ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε η Επίτροπος Τήσεων στην Ευρώπη υπάρχει μισθολογικό χάσμα 16% και συνταξιδοτικό 30% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσει κατά των γυναικών ε, και τρει φορέ περισσότερο ασχολούνται με μία βιώμενε οικιακέ εργασίε. Ε, η οδηγία περί συμφιλίωσης επαγγελματική και ιδιωτική ζωή κάνει ένα βήμα προ τα μπρο για την κοινωνική Ευρώπη για την οποία τόσο μιλάμε αλλά δεν πράττουμε γιατί αυτή η οδηγία θα επιτρέψει μία πιο ισότιμη κατανομή ε, των ευθυνών κοινών φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αποτελεί λοιπόν μια προώθηση της ε, ισότητας αλλά και αναγνωρίζει και νέα δικαιώματα όπως ε, το να ζητούνται ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για τη φροντίδα των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι μακριά βέβαια από αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Παρ' όλα αυτά αποτελεί μια πρόοδο και συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μιράντα παρακαλώ. Και για σας ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους φροντιστές και τις οικογένειες και αυτή είναι ε, η εγγύηση ε, της ισότητας ε, γιατί αποτελεί ένα βήμα προς τον τη Ευχαριστώ την δυνατότητα που δίνεται στα κράτη-μέλη να βελτιώσουν και να συμφιλίσουν την Οι γυναίκες είναι πάντα αυτές που μένουν στο σπίτι, που αφήνουν τη δουλειά τους και αυτό δεν είναι σωστό. Επίτροπε στη χώρα μου ε, υποφέρουμε από γύρανση του πληθυσμού ε, και ε, είναι τα παιδιά, συγγνώμη, είναι οι παππούδες που φροντίζουν τα παιδιά. Πρέπει να δίνουμε άδειες γονικές και θα πρέπει να φροντίζουμε τους ασθενείς και τα εξερτώμενα μέλη. Η μητέρα μου έχει Αλτσχάιμερ και αυτό μας άλλαξε τη ζωή, όπω σε τόσε οικογένειες και στη χώρα μου και σε όλη την Ευρώπη. Οι φροντιστές και οι οικογένειε χρειάζονται την υποστήριξή μα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καπούτο παρακαλώ για ένα λεπτό τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ. Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προ τα μπρο, προ μια καλύτερη ισορροπία για όλου του γονεί που εργάζονται. Έχουμε ένα ελάχιστα πρότυπα για του γονεί που μπορούν να ζητήσουν, οι πατέρε μπορούν να ζητήσουν τουλάχιστον 10 μέρε άδεια μετά τη γέννηση ενό παιδιού. Η δυνατότητα μεταφορά τη άδεια τουλάχιστον για δύο μήνε, τουλάχιστον θα πληρώνεται όπως το επίπεδο, το επίδομα ασθενείας. Ε, η άδεια για τους ε, φροντιστές ε, φτάνει τις πέντε μέρες ετησίως και όλοι οι γονείς με παιδιά κάτω των 8 ετών θα μπορούν να ζητήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία τους. Στην πράξη προσφέρεται στις οικογένειες με γονείς και ε, με παιδιά, συγγνώμη, ε, μια δυνατότητα να συμφιλιώσουν την επαγγελματική και ιδιωτική τη ζωή. Είναι ένα τεράστιο βήμα προ τα μπρο για μια νέα Ευρώπη, μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Και τώρα η κυρία Τίσεν για να απαντήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, όπως ξέρετε, και ορισμένοι το αναφέρατε κάτι στη συζήτηση, η διαπραγμάτευση δεν ήταν εύκολη. Και έχουμε κάνει όλοι μεγάλες προσπάθειες ε, και όλοι χρειάζεται να δείξουμε διάθεση συμβιβασμού για να επιτύχουμε ορισμένα θέματα, αλλά θεωρώ ότι η συμφωνία που έχουμε ενώπιόν μας είναι ισορροπημένη και διατηρεί τους βασικούς στόχους αρχικής μας πρότασης. Αποδεικνύει ότι η κοινωνική Ευρώπη και η βιώσιμη Ευρώπη δεν είναι ένας ε, ανέφικτος στόχος, αλλά μια απτή πραγματικότητα. Είμαι πεπισμένη ότι θα βελτιωθεί σαφώς και συγκεκριμένα η οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των ε, συμπολιτών μας και θα κάνει τον κοινωνικό πυλώνα πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο θέμα ε, δικαιοσύνης, αλλά ωφελεί τους πάντες και τους εργαζόμενους γονείς και αυτούς που παρέχουν φροντίδα θα έχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού είναι καλό και για τις επιχειρήσεις και μάλιστα τις μικρομεσαίες που θα μπορούν να προσελκύουν και να διατηρούν ταλαντούχους εργαζόμενους και θα είναι καλό για τα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή χάνουν 370 δισεκατομμύρια λόγω του χάσματος ε, στη σχέση, στην ε, ίση μεταχείριση των φίλων. Θεωρώ ότι η οικογενειακή ζωή είναι βασικός παράγον για την οικονομική ανάπτυξη. Σας καλώ λοιπόν όλους να στηρίξετε την οδηγία για την ισορροπία επαγγελματική και προσωπικής ζωής Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προ εμένα προσωπικά. Και σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά την μεταφορά τη οδηγία αυτή στο Εθνικό Δίκαιο. Σε ευχαριστώ πολύ για τους κόπους σας και την αφοσίωσή σας για αυτό το θαυμάσιο έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα φυσικά τελευταίος ο εισηγητής, Ντάβιτ Κάζα. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την, Επιτροπο, την αλλά και την κυρία Γιώργοβα για την πολύτιμη βοήθεια και υπομονή που έδειξαν σε, τη, όλη τη διάρκεια των συνομιλιών τη συνάδελφο Αγνιέσκα αλλά και όλους τους ε, σκιώδεις συγκητές που συνεργάστηκαν μαζί μου στην οδηγία αυτή. Κάποιοι σκιώδεις δεν έδειξαν καμία διάθεση συνεργασίας. Κάποιοι διεκδικούσαν πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε να προσφέρουμε. Ωστόσο, θα ακούσατε όλοι σήμερα πως οι περισσότεροι σκιώδεις συμφώνησαν πως πρόκειται για μια λύση νομοθετική ισορροπημένη και από τις συζητήσεις που είχαμε και με την Γενική Συνομοσπονδία των Εργασμών στην Ευρώπη και με άλλες ομοσπονδίες ε, είδαμε πως μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό δηλαδή το οποίο προτείνουμε σήμερα με την οδηγία αυτή εξασφαλίζει μια Ευρώπη περισσότερο κοινωνική από ότι σήμερα. Και έτσι δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συζήτηση που έγινε σήμερα, η οποία και αντικατοπτρίζει και Τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο αλλά και τι συνομιλίε με το Συμβούλιο οι οποίες αρχικά είχαν ε, αρκετέ δυσκολίε. Με τον καιρό όμω είδαμε πως αρκετά μέλη του Συμβουλίου, τα περισσότερα ήταν υπέρ των προτάσεων και έτσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε μαζί. Δεν είναι κάτι το οποίο επέτυχε ένας άνθρωπος μόνο του το αποτέλεσμα που βλέπετε. Πρόκειται για τον καρπό της συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και καταλήγω λέγοντας πως πρόκειται για, μια, για ένα νομοθέτημα καλό, εξισορροπημένο για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες για την οικονομία πάνω απ' όλα όμως ένα καλό για την κοινωνική Ευρώπη νομοθέτημα. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές όσοι έλαβαν το, όσο έλαβαν λόγο, την Επίτροπο που είναι ακόμη εδώ και διακόπτω προς το παρόν μέχρι τις 11 και τις ψηφοφορίες.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

καλά να Präsident! Die Sitzung Αρχίζει η συνεδρίαση. Εχθέ η Ολομέλεια ενημερώθηκε ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ δεν σκοπεύει να εγείρει αντιρρήσει σε κατεξουδότηξη πράξη και έτσι οι συστάσει δυνάμει του άρθρου 105.6 θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί, δημοσιεύονται δε μαζί με τα ε, υιοθετηθέντα έγγραφα. Παρακαλώ να λάβετε τι θέσει σα για να περάσουμε στι ψηφοφορίε. Και ξεκινώ με την έκθεση Τσαμπάτσκι. Πρόταση απόφασης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν την άρση ασυλίας μου γιατί μετά τη δολοφονία του γιού μου Γιώργου Φουντούλη από τρομοκράτες παραμένουν ασύλληπτοι. Μετά από δεκάδες επιθέσεις και καταστροφές στα γραφεία μας με εκρηκτικούς και εμπριστικούς μηχανισμούς από παρακρατικούς της αριστεράς και την αδιαφορία της ελληνικής αστυνομίας να μας προστατεύσει κάναμε το τεράστιο έγκλημα να τοποθετήσουμε κάμερες ασφαλείας για να προστατεύσουμε Πρόεδρος, δεν είχαμε προβλέψει να γίνει συζήτηση πριν από την ψηφοφορία για τις ασυλίες, κύριε συνάδελφε και ως εκ τούτου δεν μπορώ να σας επιτρέψω να συνεχίσετε την τοποθέτησή σας. Συνεχίζω λοιπόν με την έκθεση Τσαμπάτσκι. Υπέρ, κατά, αποχές και εγκρίνεται Άλλη μια έκθεση Σαββάτσκι. Ασυλία του κυρίου Συναδεινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. Φόξ. Πρόεδρε, επικαλούμε το 194. 90 παράγραφο. 44. Θα ήθελα να παραταθεί το θέμα το θέμα αυτό για την επόμενη σύνοδο γιατί δεν είναι δυνατόν να περιγράφεται στο σχετικό, στη σχετική έκθεση η, για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τη θεώρηση η, το Γιβραλτάρ ως απικία. Είναι ε, ένα έδαφος, μια εδαφική οντότητα η οποία επέλεξε να ενταχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης 59 ψήφοι υπέρ με μηδέν κατά ήταν αυτές που έδωσαν από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών την εντολή στον Κλοντ Μωράες ο οποίος έκανε τη δουλειά του ε, βαζόμενος σε αυτή την την εντολή, ωστόσο ε, του αφαιρέθηκε η εντολή επειδή οι επιλογές του δεν, δεν βρήκαν σύμφωνους εκείνους οι οποίοι παραβιάζοντας την, ε, τον κανονισμό αφαίρεσαν την έκθεση από τον κύριο Μωράης. Άλλο να έχουμε κάποιες θέσεις για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλο να παραβιάζουμε τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν να γίνει συζήτηση για να καταγγελθεί η διεφθαρμένη ε, στάση που έχει τηρήσει η Ισπανία στην υπόθεση αυτή. Πρόεδρος, 190 παράγραφος 4 λοιπόν, εναντίον της πρώτης κυρία Γκαρσία Πέρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν θα επιτρέψω να προσβάλλετε την κυβέρνηση της Ισπανίας, γιατί πρόκειται για προσβολή απέναντι στην πλειοψηφία των πολιτών της χώρας μου. Δεύτερον, δεν γίνεται οι δημοκρατικές διαδικασίες να τις συνδετούμε όταν είναι υπέρ μας. Εδώ είχαμε μια διαδικασία συμφωνίας με το Συμβούλιο, όπως συμβαίνει και σε πολλά άλλα ζητήματα όπου το Συμβούλιο έθεσε τη θέση του, το Κοινοβούλιο τη δική του και υπήρξε διαπραγμάτευση όλη η διαδικασία και η λήψη απόφασης έγινε σύμφωνα με τον νόμο, έτσι όπως ε, θεσπίζεται. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ επικύρωσε την αλλαγή του εισηγητή και επομένως πρέπει να δεχτείτε την απόφαση αυτή. Και τέλος, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτοί που θα αποχωρήσουν να αποφασίσουν επί των συμφερόντων όσων μένουν. Στην συμφωνία ορίστηκε ένας ορισμός που συνάδει με το διεθνές δίκαιο και να μην ξεχνάμε, εδώ αυτό που ψηφίζουμε σήμερα δεν αποτελεί συνέπεια μιας απόφασης της κυβέρνησης της Ισπανίας. Εδώ σήμερα ψηφίζουμε ότι αν στις 12 Απριλίου αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει επιληθεί το θέμα της απαλλαγής από τις θεωρήσεις. Και κόβετε το μικρόφωνο της ομιλίας. Ευχαριστώ κυρία Γκαρθία Πέρεθ. Λοιπόν, ε, ποιο είναι υπέρ του να αναβληθεί ζήτηση για το θέμα αυτό. Ποιοι είναι κατά. Λοιπόν, καλά, καλά, θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο τώρα. Η κυρία Γκέρλινγκ, παρακαλώ, ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Για το ίδιο θέμα, αλλά με βάση το 59.3 άρθρο του στροκονισμού. Καλό την, ε, το σώμα να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε την έκθεση. Δεν θέλω να αναβληθεί. Είναι τεχνική και ιδιαίτερα καλοδεχούμενη έκθεση που δίνει δυνατότητα οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου να μπαίνουν στην Ένωση. Στην ουσία έχει αλλάξει χαρακτήρα λόγω της, ε, για πολιτικούς λόγους στάσης ε, της κυβέρνησης Ισπανίας στο Συμβούλιο. Να περιγράφεται ως ε, απικία το Γιβραλτάρ δεν ήταν στην διαπραγματική εντολή του Κοινοβουλίου και ο εισηγητής Μωράης πάντα στήριξε την άποψη του Κοινοβουλίου. Υπέστη τρομερές πιέσεις και τελικά του αφαιρέθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων η έκθεση αυτή και κατόπιν το Κοινοβούλιο πολύ ταχαίως δέχτηκε τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου. Στην ουσία είναι συνέργεια του Κοινοβουλίου για να αντικατασταθεί ένα κείμενο που νόμιμα είχε ε, αποφασιστεί από το Κοινοβούλιο για λόγους ίδιου συμφέροντος ενός κράτους μέλους. Ανεξάρτητα από την πολιτική φύση, νομίζω ότι αυτό είναι σωστή παραβίαση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εγώ και 38 ε, συνάδελφοι, διακόπτει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Γκέρλινγκ. Πρώτα απ' όλα το θέμα αν υπάρχουν 38 συνάδελφοι ε, που συμφωνούν με αυτό το αίτημα. Νομίζω ότι υπάρχουν. Υπάρχει αφιβολία. Υπάρχει καμία αφιβολία. Ποιο θέλει να μιλήσει κατά του αιτήματο αυτού. Ο Σάλβος Γκονθάλεφ Πόνς. Κύριε Πρόεδρε. Μη φοβάστε. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που ψηφίζουμε τώρα εδώ είναι η εξαίρεση για προξενικές θεωρήσεις για εκατομμύρια πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν την επόμενη εβδομάδα γίνει σκληρό Brexit. Εάν αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία, αν τροποποιήσουμε την έκθεση, σημαίνει ότι θα καταδικάσουμε εκατομμύρια Ευρωπαίους να πρέπει να ζητήσουν βίζα για να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, για λόγους ιδίου συμφέροντος της Βρετανικής κυβέρνησης θέτουμε κινδύνο τα ταξίδια εκατομμυρίων πολιτών. Άρα δεν μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία ούτε να δεχθούμε τροπολογίες. Λυπάμαι. Οι Βρετανοί θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καθήκον μα είναι να προστατεύσουμε του συμπολίτε μα. Και αυτό σα ζητώ να κάνουμε τώρα. Αυτό ζητώ από το σώμα να κάνει. Λοιπόν, να ψηφίσουμε, λέει ο πρόεδρο. Ποιοι ε, είναι υπέρ τη πρόταση κυρία Γκέρλινγκ, παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Καλά να το ελέγξουμε και αυτό. Καλά μην εκνευρίζεστε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Οπότε, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την προσωπική συμφωνία ε, τροπολογία 3 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην έκθεση Μητροφάνοφς. Προφορική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Τώρα έχουμε τη διαχείριση των αποβλήτων. Ε, ψήφισμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Οπότε, έκθεση κιλών. Αγαπητή. Λοιπόν, θα κάνουμε πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Σήμερα το πρωί έλαβα πολλά τηλεφωνήματα. Σας είδα, σας είδα για αυτή την ψηφοφορία, σας είδα. Σας διαβεβαιώ ότι ήρθα με το αυτοκίνητο, ε, θα φύγω αύριο, έχω όλο το χρόνο στη διάθεσή μου. Επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μέσω του κανονισμού να γίνουν ψηφοφορίες ε, με μπλοκ ψηφοφοριών. Αλλά φυσικά οι υπηρεσίες θα καθορίσουν, θα προετοιμάσουν αυτές τις ε, αυτά τα μπλοκ. Ξέρω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικέ απόψει για αυτά, οπότε θα πρότεινα στην αρχή να αρχίσουμε την ψηφοφορία και μετά από λίγο χρόνο θα σας ρωτήσω εάν πραγματικά θέλετε να ψηφίσετε κάθε μεμονωμένη τροπολογία ή, θα ή αν θα μπορούσαμε να κάνουμε ψηφοφορία σε μπλοκ. Διαδικαστικό εσείς παρακαλώ κύριε. Η κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το θέμα δεν είναι ο χρόνος. Το θέμα είναι να έχουμε ένα καλό νομοθέτημα μετά την ψηφοφορία. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ότι έχουν ομαδοποιηθεί οι τροπολογίες με τα ονόματα των συντακτών των τροπολογιών. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το νομοθέτημα που θα προκύψει δεν θα είναι καλό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις θέσεις εργασίας και εμείς θα γίνουμε περίγελος. Έτσι λοιπόν ζητάμε έναν κατάλογο ψηφοφοριών που να έχει προετοιμαστεί σωστά. Έχουμε 1.400 τροπολογίες, θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε έναν κατάλογο ψηφοφοριών για το Στρασβούργο. Έτσι λοιπόν απευθύνω έκκληση σε όλους να υποστηρίξετε το αίτημα αυτό. από πλευρά ομάδας ECR προτείνω να αναβληθεί η ψηφοφορία αυτή γιατί η αλληλουχία των τροπολογιών παραβιάζει το 174.2 και 8 του εσωτερικού μας κανονισμού. Ε, υπάρχουν δύο εναλλακτικέ λύσεις έχουμε ταυτόσιμες τροπολογίες που είναι σε διαφορετικά μπλοκ και θα, αν το ψηφίσουμε έτσι δεν τηρούμε το 194-9 του ιστορικού κανονισμού. Έχουμε βρει τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις γιατί αυτά τα μπλοκ τροπολογιών έχουν συσταθεί με βάση τους συντάκτες των τροπολογιών και όχι με βάση το περιεχόμενο των τροπολογιών. Και αυτό είναι απόλυτα αντίθετο με μια σωστή διαδικασία. Οπότε, Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μέσα αυτή τη διαδικασία να κάνουμε σοβαρό διαδικαστικό λάθο και μπορεί γι' αυτό να γίνουν προσφυγέ στα δικαστήρια. Για τρίτη φορά κατά την τρέχουσα θητεία. Οπότε κάνω έκκληση να στηρίξετε το αίτημά μου για αναβολή. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Πολύ ευχαριστώ. Εάν όμως είχατε την καλοσύνη, αντί να διαβάζετε έτοιμες από πριν ομιλίες, να ακούγατε τι έχω πει, δηλαδή ότι πρόκειται να ψηφιστεί αυτό το αίτημα. Η κυρία πριν από εσά έκανε το ίδιο αίτημα για αναβολή και ως εκ τούτου, χωρίς να θέλω να ε, επιμείνω περισσότερο, θα προτείνω να ψηφίσουμε τώρα. Ψηφίσαμε και χτες. Άλλη μια φορά τώρα λοιπόν. Υπέρ της αναβολής παρακαλώ υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Εξακόσια παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 630 όχι ζητώ συγγνώμη 645, 691, 650 και λοιπές τροπολογίες που προτείνουν την απόρριψη ονομαστικά. Παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρασε. απερίφθησαν. Και έτσι πάω στην 629 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 630 Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε πολύ καλά ότι μετά γίνεται το αίτημα για την επαλήθευση. Θα κάνω ό,τι μπορώ σήμερα για να φυλάξω ομαλέ κοινοβουλευτικέ διαδικασίε, αλλά δεν θα επιτρέψω και σε κανένα να παρεμποδίσει τι ψηφοφορίε. Και παρακαλώ να μην υπερβάλλετε. Deshalb lasse ich das jetzt zunächst mal überprüfen. Άρα κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται παρακαλώ η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε. Πέρασε ψηφοφορίας απορρίπτεται και χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων να το έχετε αυτό υπόψη βέβαια είναι ξεκάθαρο ε, το αποτέλεσμα δεν θα ζητώ πάλι 6.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εντάξει ελέγχουμε την 630 άρχεται η ψηφοφορία alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 631 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 632. Να ελέγξουμε την 631. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφεται και εδώ με την πλειοψηφία των δύο τρίτων. Θέλετε το λόγο τη διαδικασία. Ναι. Για διαδικαστικό ήθελα το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο και θα πρότεινα να συνεχίσουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, δυνατόν. Με επιτρέπετε κυρία Γκραπή να το αποφασίζω εγώ αυτό. 633 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 633 λέω τώρα πρόεδρος. 634 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 635 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 618 ψήφι υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται 619 ψήφι περ. Κατά αποχές απορρίπτεται 620 ψήφι περ. Κατά αποχές απορρίπτεται 621 ψήφι περ. Κατά αποχές απορρίπτεται 622 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 623 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 624 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 625 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 626 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 627 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 628 ψήφι περ. Κατά αποχές απορρίπτεται 636 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 637 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 638 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 631 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 640 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 641 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 642 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 643 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 644 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ολοκληρώσαμε την πρώτη δέσμη, αγαπητοί συνάδελφοι. 1100 συνολικά αντροπολογίε. Περνάμε στην δέσμη Β. Και προχωρούμε 763 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 292 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 293 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 294 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 295 με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 296 με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. abgestimmt η Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 207 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.98 ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.99 ψήφι περ. Κατά αποχές απορρίπτεται 300 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 301 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές απορρίπτεται 302 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές απορρίπτεται 303 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 304 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 224 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται 225 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 226 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 227 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 228 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 229 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 230 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 231 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 232 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 2.33 ψήφι πέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 2.34 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται 2.35 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.36 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.38 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.39 ψήφι πέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2.40 ψήφι κατά αποχές το 2.41 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.42 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.43 ψήφι υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 2.44 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.45 ψήφι υπέρ κατά αποχές από το 246 ψήφι υπέρ κατά αποχές από το 247 ψήφι υπέρ κατά αποχές από απορρίπτεται 248 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται 249 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 250 ψήφι πέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 251 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 252 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 253 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 254 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 255 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 256 ψήφι υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 257. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 258. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 259. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 260. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δεν μπορώ να πάω πιο γρήγορα, δεν μπορείτε ούτε εσείς πιο γρήγορα, ούτε και οι διερμηνείς μπορούν πιο γρήγορα. Και επειδή έτσι όπως παρατηρώ τελευταία ε, υπάρχουν πολλές, πολύ μεγάλη διαφορά από 550 έως 2 τρίτα ψηφίστε υπέρ συνήθως, οπότε το σκέφτομαι μήπως τελικά ε, να ακολουθήσω την ε, υπόδειξή σας να ψηφίσουμε ομού. Lassen Ας δώσουμε δύο-τρία λεφτά στο να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Κύριε Μαρινέσκου. Dear colleague, dear Vice President. Κύριε Αντιπρόεδρε, άκουσα το αίτημα των συναδέλφων από την αρχή, αλλά αυτό που ψηφίζουμε δεν αφορά το περιεχόμενο αφορά περιφερεια... τα... την αντιπαράθεση της περιφέρειας σε σχέση με, την... με τον πυρήνα. Άρα, ας ψηφίσουμε άρθρο προς άρθρο, παράγραφο προς παράγραφο, στο περιεχόμενο δηλαδή. Γιατί δεν πρέπει να ψηφίζει έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να ψηφίσουμε ανά ομάδες ε, τροπολογιών είναι ότι υπάρχουν ομάδες βουλευτών που πρότειναν τροπολογίες. Σε ένα μπλοκ υπάρχει, ας πούμε, τροπολογία για το άρθρο 4, 9, 12, που είναι άσχετες μεταξύ τους. Απ' τη μία μιλάμε για την, το χρόνο οδήγησης, για την ηλικία του οδηγού, για το που παρκάρει το φορτηγό του κτλ. Καμία σχέση. Άσχετες τροπολογίες δηλαδή θα, θα ψηφίσουμε μαζί. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν ακολουθούμε τους κανόνες του Κοινοβουλίου. Φταίνε οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου για αυτό το χαμό που δημιουργήθηκε. Κύριε Μαρινέσκου, όλα αυτά που είπατε τα ακούω αλλά ε, αποκρούω αποφασιστικά την τελευταία σας πρόταση. Ε, κύριος Λαμπέρτς, ε, Πρόεδρε, ακούω αυτό που λέει ο κύριος Μαρινέσκου ότι ομαδοποιήσαμε βάσει των συντακτών της ε, Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά ακριβώς οι ομάδες των τροπολογιών έχουν μια πολιτική λογική. Δηλαδή, οι διάφορες ομάδες των συντακτών των τροπολογιών το έκαναν έχοντας μια καθολική εικόνα το άρθρο και μάλλον την, ε, της έκθεσης βέβαια σε διάφορα άρθρα αλλά έχουν ε, πολιτική συνάφεια και συνοχή μεταξύ τους συντροπολογίες οπότε έχει νόημα να τις ψηφίσουμε ομαδών. Ωραία. Ακούσαμε τις δύο απόψεις. Προσωπικά ε, θεωρώ κύριε Μαρινέσκου ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να γελιοποιείται και από διάφορες κατευθύνσεις. Μπορούμε να γελιοποιηθούμε και ψηφίζοντας σαν μπλοκ, αλλά και ε, ακολουθώντας τη διαδικασία που ε, ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Το θέμα είναι να βρούμε μια αντικειμενική λύση που να εξυπηρετεί το σκοπό μας. Έχουν γίνει κάποιες προεργασίες ε, στην Επιτροπή, την Αρμόδια, που πρέπει να ληφθούν και αυτές υπόψη και τίνω να συμφωνήσω περισσότερο με τον συνάδελφο Λάμπερτς. Και σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού έχουμε τη δυνατότητα να ομαδοποιούμε τις τροπολογίες και υπάρχει και αποχρό λόγο γι' αυτό. Και θα δώσω λόγο στον κύριο Κόρμπετ που φέρει και την κύρια ευθύνη του κανονισμού. Yes, Ομολογώ, Πρόεδρε, εγώ, ότι εγώ συνέταξα αυτή την παραγραφό του εσωτερικό κανονισμό και υπάρχει εδώ και χρόνια αυτή η διάταξη. Υπάρχει ακριβώς για να προβλέψει τέτοιες καταστάσεις όπου έχουμε ασυνήθιστο αριθμό τροπολογιών και μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις τροπολογίες όπως ακριβώς περιέγραψε ο κύριος Λάμπερτς ή με άλλους τρόπους, με λογικό πάντα τρόπο ούτω ώστε να μπορέσει να εργαστεί σωστά το Κοινοβούλιο με σεβασμό των απόψεων των βουλευτών. Έχει νόημα να ομαδοποιήσουμε τις τροπολογίες με αυτόν τον τρόπο και θα μας επιτρέψει να εργαστούμε αποτελεσματικά χωρίς να χάσει κανένας βουλευτής το δικαίωμά του να υποβάλει τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Κόρμπετ. Λοιπόν, δεν θα δώσω το λόγο τώρα για διαδικαστικό και επί του κανονισμού σε κανέναν. Ακούσαμε δύο απόψεις και μία εξήγηση. Θα μπορούσα να το αποφασίσω μόνος μου και ε, άφησα να νεωθεί ότι συμφωνώ με τον κύριο Λαμπέρτς, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εσάς, συμφωνείτε να ψηφίσουμε ομαδικά τώρα τις τροπολογίες, μπλοκ, ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Das lasse ich überprüfen. Die... Ας το ελέγξουμε παρακαλώ, άρχεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Haben alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Με πλειοψηφία δύο τρίτων, αν είναι σωστή υπολογιστή μου. Άρα, το μπλοκ Β, λοιπόν, συνεχίζουμε από την 261 μέχρι ε, την 332. Ε, Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ, αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση του μπλοκ αυτού. Ψηφίσατε όλοι. Die Abstimmung geschlossen abgelehnt mit annähernd zwei Drittel Mehrheit. Block ε, απορρίπτεται. Το μπλοκ ε, Γ, C, υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. D. Der Kollege hinten hat sich zuerst ο συνάδελφο πίσω ζήτησε το λόγο ε, επί του κανονισμού. Σε ποιο άρθρο αναφέρεστε παρακαλώ. Πρόεδρε, γιατί θα ψηφίσουμε έτσι. Εγώ διαφωνώ στις διάφορε τροπολογίες. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω υπέρ ή κατά. Υπάρχουν τροπολογίες στα μπλοκ που υπερψηφίζω και άλλες καταψηφίζω. Αυτό είναι παρεμπόδιση και παρακόλληση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του δικαιώματος άσκηση ε, άσκησης ελευθερία της ελευθερίας του βουλευτή. Ο κύριος Γιούρεκ. Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα την ιδέα του να ψηφίσουμε ομαδικά τις τροπολογίες. Αλλά εφόσον το αποφασίσαμε και αν υπάρχουν ονομαστικές ψηφοφορίες εντός του μπλοκ, τότε θα πρέπει να ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση όλο το μπλοκ, αυτό, όλη την ομάδα αυτή των τροπολογιών. Έτσι, με ονομαστική κλίση. Κύριε Γιούρεκ, και γιατί δεν μαρτύρεστε, δεν καταλαβαίνω. Μέχρι τώρα δεν ψηφίσαμε κανένα μπλοκ που να ζητούσε ονομαστική ψηφοφορία και ακριβώς αυτό θα σας πρότεινα τώρα το μπλοκ D να το ψηφίσουμε συνολικά ονομαστικά και αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Abgelehnt. Απορρίπτεται. Μπλοκ ε έχει επίση ονομαστική, άρα ψηφίζουμε ολόκληρο το μπλοκ ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και αν ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μπλοκ F. Ονομαστικά και αυτό αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία.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 τα block H έως K ε, καταπίπτουν. Συνολική ψηφοφορία τελική, ονομαστική και αρχίζει τώρα παρακαλώ.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 Θα ήθελα να σας πω ότι και το Block G διεκπαιρεώθηκε και κατέπεσε εφόσον εγκρίθηκε προηγούμενο. Πάμε τώρα στην έκθεση Κάμπ. 307 και 423 ονομαστικά ταυτίζονται αυτές οι δύο τροπολογίες. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Διαφωνείτε να ψηφίσουμε πάλι έτσι με μπλοκ τις τροπολογίες. Ο κύριος συνάδελφος Ευχαριστώ. Θα υπήρχε η δυνατότητα, μια που θα ψηφίσουμε unblock, να κάνουμε όλες τις, ε, τις ψηφοφορίες ηλεκτρονικά. Όχι μόνο εκεί που λέει ονομαστική, να τις κάνουμε όλες ηλεκτρονικά από την αρχή. Βεβαίω, με χαρά, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, το πρώτο μπλοκ. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το δεύτερο μπλοκ. Ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, όχι. Τώρα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το τρίτο μπλοκ, C. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μπλοκ D. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μπλοκ ε. Άρχιτη η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. F ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, ε τα μπλοκ G και H τώρα καταπίπτουν και θα ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά. Αρχίζει τώρα παρακαλώ η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση Ερτούγκ. Οι τροπολογίες 290 και 308 είναι ταυτόσιμες. Αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. Απορρίψετε. Το μπλοκ Α. Ο κύριος Στεχόφσκι ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε, για το άρθρο 182α. Είμαι κατά. Είμαι κατά του τρόπου που διενεργείται την ψηφοφορία. Για λόγους που θα υποβάλω γραπτός στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι παραβιάζονται διάφοροι κανόνες με τον τρόπο που δουλεύουμε. Διάφορα σημεία του εσωτερικού κανονισμού. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό το πρόβλημά μου. Ευχαριστώ, το λαμβάνω υπόψη. Μπλοκ Α, ονομαστικά, ε, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Πέρασε. Μπλοκ Β, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Haben alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μπλοκ C. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μπλοκ D. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Μπλοκ ε, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Άρα τα μπλοκ F και G εμ, καταπίπτουν και ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία. Τελική είναι αυτή. Μάλιστα. Ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Die Abstimmung ist geschlossen. sind bei allen drei Berichten Οπότε ολοκληρώθηκαν οι αναγνώσεις και για τις τρεις εκθέσεις που ψηφίσαμε. Έκθεση Μπούζεκ, προσωρινή συμφωνία, είναι η τροπολογία 23, ονομαστικά ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. angenommen. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στην έκθεση ΜΑΤΟ τι ε, τροπολογίε ε, τη Αορμάς Επιτροπής υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνονται. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 18 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 σε 3 τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 τροπολογία ψήφι υπέρ, κατά, αποχές... Νομίζω απορρίπτεται, ας το ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία για την 37. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. τροπολογία 38 ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. Τροπολογία 44 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 48 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 50 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 53 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 54 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 80 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 93 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 116 ψήφι υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται 117 ψήφι υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 120 ψήφι υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 121 ψήφι υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 123 ψήφι υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 126 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 138 με ονομαστική και αυτή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. 141 ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται 152 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 156 μονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 157 μονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται 158 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 159 ψηφιπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 165 ψηφιπέρ κατά, απόχέ εγκρίνεται. 168 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 171 ψήφι υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 178 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 182 ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται 188 ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται 190 ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται 195 ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται 196 ψήφι περ κατά αποχές θα ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία 196 ψηφίσατε όλοι Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 198 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 200 ψήφι πέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 205 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 224 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 259 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 264 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 268 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 269 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 270 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 274 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 275 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 291 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 84 λοιπόν κατά 291 CP2. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται κατά 86. 281 ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουν παρακαλώ, έχετε ψηφοφορία. Και καλό θα ήταν ε, να παρακολουθείτε καλύτερα αυτούς που δείχνουν ότι πρέπει να ψήσετε είναι, και αυτή είναι η πιο ορατή. Εγκρίθηκε. 2.92 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. περαση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 90. Ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92. Ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 293 κατά 282 τώρα ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές εγκρίνεται άρα 314 όχι εντάξει ελέγχουμε ελέγχουμε την 282 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 3-14 ψήφι υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά κάπως ε, ε, μετακινήστε ως προς το, στις ψήφους σας και δεν μπορώ να καταλάβω άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Απορρίπτεται το 94 τώρα Περκατά κατά αποχές εγκρίνεται. 283 και 315. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ελέγχουμε. 283 και 315 ταυτόσιμες τροπολογίες άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen εγκρίνονται. 34 και 95 καταπίπτει και 95. Ναι. Άρα πηγαίνουμε στην 96. 96 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 96 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα, κατά πίπ 316, 317 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα 100... ελέγχουμε την 317 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει 113-284 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο του άρθρου 13 παράγραφος 1 σημείο β πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 13 1 δέλτα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 1 ε ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 1 μάλλον 124 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατα το αρχικό πίπτου 13.1. Πάμε στο 13.1J, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. Να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κατά πριν αρχικό κείμενο. 323 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 310 ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται 311 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 322 ψήφι πέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 135 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απορρίπτεται 285 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ έχει νόημα όχι έχει υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 318 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 312 τροπολογία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας Εγκρίνεται. 16.3α αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.86 ψήφι ΠΕΡ. Κατά αποχές απορρίπτεται 142 ψήφι ΠΕΡ. Κα, ε, κατά αποχές Ελέγχουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 142. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Άρα το αρχικό κείμενο ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 144 ψήφι πέρα κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται αρχικό κείμενο με ονομαστική. Α, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. 155 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. εγκρίνεται. 3.13 και 3.20 καταπίπτουν αρχικό κείμενο 18.4 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Abgelehnt. Απορρίπτεται. 321 ε, υπέ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.19 είπε. Α, όχι, εντάξει, έχει καλυφθεί. Και οι 2.49 και οι 300 ε, ονομαστικά είναι ταυτόσιμες αυτές. Ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ. Εγκρίνονται. 287 ψηφίπε κατά αποχές εγκρίνεται Άρα η 221 καταπίπτει, 302 σε δύο τμήματα, ονομαστικά τμήμα πρώτον, άρχη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και το δεύτερο τμήμα δεν έχει νόημα να το ψηφίσουμε. 217 και 301 ονομαστικά οι δύο αυτές ταυτόσημες. Άρχισε ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνονται. 303 ονομαστικά άρχη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 έχει καλυφθεί. 277 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 288 και 9 ναι, καταπίπτουν 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 καταπίπτει θέλετε έλεγχο για τη 278 παρακαλώ άρχιτε ψηφοφορία Εάν ψηφίσατε όλοι Πέρασε. απορρίπτεται. Η 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 289 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 304 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 279 υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. Και καταπίπτει 32. Θέλετε έλεγχο για τη 279, παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 32, 305 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται οι 40 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές μάλλον έχει εγκριθεί αλλά στο επαληθεύσουμε 306 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 307 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 290 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 280 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 309 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το σύνολο της πρότασης, όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά, Αρχίζει η ψηφοφορία. Αν ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται ούτω λοιπόν η πρώτη ανάγνωση. Έκθεση Αγγιλέρα Γκαρθία. Ε, προσωρινή συμφωνία, τροπολογία 97, ονομαστική κλίση, αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η κυρία Καλνιέτε, επί του κανονισμού. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ψηφίσαμε και δαπανίσαμε πολύ περισσότερο χρόνο για το κείμενο του ΜΑΤΟ παρά για το πακέτο κινητικότητας. Κυρία συνάδελφε, κυρία Καλνιέτε, δεν μου διέφυγε. Η τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην έκθεση ΔΕΠΧΕ τώρα. Η κυρία Έρνστ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ, η κυρία Έρνστ. Με μικρόφωνο. Παρακαλώ, βάσει ε, του άρθρου 59 του κανονισμού, να ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες. Θέλει να διαφωνήσει κανείς με το αίτημα αυτό. Όχι από ό,τι βλέπω. Ο εισηγητή ζητεί το λόγο. Κύριε Ντεπρέ, παρακαλώ. Ε, Ω εισηγητή, ζητάω από, τις, ε, από τους συναδέλφους να απορρίψουν τις προτάσεις της ΓΚΟΕ. Η συμφωνία είναι καρπός διαπραγματεύσεων και είναι πολύ ισορροπημένο ε, διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Και η υιοθέτηση σε, μία τροπολογία της θα, θα καθιστούσε τη συμφωνία με το Συμβούλιο ε, άκυρη. Κάτι που θα ήταν πολύ ε, μεγάλο πρόβλημα για την ελεύθερη κυκλοφορία και την ταυτότητα. Και τις πλαστές ταυτότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ονομαστική ψηφοφορία το αίτημα της κυρίας Σέανς θα αρχίζει τώρα, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Die Abstimmung ist geschlossen. Απορρίπτεται. Άρα, και οι τεχνικοί έχουν πολύ δύσκολη δουλειά, όσο και όλοι οι υπόλοιποι. Και μην εκνευρίζεστε αν διαρκεί λίγο παραπάνω ε, το να ανοίξει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την προπο... Ε, προσωρινή συμφωνία, συγγνώμη, 73 ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Αγιούτο. Η τροπολογία 66 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση Νιτβέλτ. Η τροπολογία 2 ονομαστικά αρχίζει τώρα. Η ψηφοφορία. Alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 3, η προσωρινή συμφωνία και πάλι ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η πρώτη ανάγνωση του κοινοβουλίου ολοκληρώνεται ούτως. Έκθεση Κάζα. Η κυρία Γκονζάλεθ Πένια ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με βάση το άρθρο 59 θα θέλαμε να ψηφίσουμε καταρχήν τις τροπολογίες. Νομίζουμε ότι είναι εκ των όνου το Κοινοβούλιο να πάρει θέση πάνω σε αυτά τα θέματα ε, για τις τροπολογίες. Ε, ένα είναι η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων ε, για να υπάρχει ισότητα και εμείς οι γυναίκες να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και το άλλο θέμα είναι οι απολαβές. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, ούτως ώστε τα άτομα τα οποία έχουν παιδιά, μητέρες, πατέρες και φροντιστές, να μην πέφτουν σε κατάσταση ένδυας. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλει να μιλήσει κανείς κατά της, ε, του αιτήματο αυτού. Ο εισηγητής, ο κ. Κάζα, παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν συμφωνώ να ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες. Έχουμε μια πολύ ισορροπημένη πρόταση οι τροπολογίε θα αλλάξουν αυτή την ισορροπία. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να καταψηφίσουμε το να ψηφίσουμε πρώτα τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάζα. Ψηφίζουμε τώρα το αίτημα της κυρίας Κονσάλεθ Πένιας. Ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Ψηφίσατε όλοι. Ε, πέρασε abgelehnt. Dann kommen wir zu dem Änderungsantrag 102. Ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Angenommen. Die erste... Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται λοιπόν η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και ερχόμαστε στην έκθεση Γκαρδία Σάμπα Ρουμπία και Σαβαρμά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση της κυρίας Λόπε Φοντανιέ. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση. Έκθεση της κυρίας Σουίνμπερν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ονομαστικά αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται, ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση, έκθεση Σιλικιώτη, προσωρινή συμφωνία, τροπολογία 2, ονομαστικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, έκθεση αφρόντε και εδώ έχουμε προσωρινή συμφωνία. Η τροπολογία 42 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, έκθεση κυρίου Ρικέ, προσωρινή συμφωνία, η τροπολογία 34, ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση. Έκθεση Πιοτρόφσκι Εδώ έχουμε τις τροπολογίες 2, 3 και 4 ταυτόσημες. Ονομαστικά τις ψηφίζουμε τώρα. Αν ε, ψήφισαν όλοι, πέρας. απορρίπτονται. Η τροπολογία παριθμένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε, ολοκληρώθηκε έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση φαγιών. Ζήτησε το λόγο η συγγήτρια. Παρακαλώ, κύριε Φαγιάν. Συνάδελφοι, ο χώρος Σέγγεν είναι ένας από τους πιο σημαντικού, ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα πιο απτά. Έχει πολυάριθμα ωφέλη για του Ευρωπαίου πολίτε και τι εταιρείε. Επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών. Λόγω των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και που ξεπέρασε τα περισσότερα, τα περασμένα κράτη-μέλη, ε, τα, τελευταία χρόνια, συγγνώμη, έξι κράτη-μέλη επί τρία χρόνια και μάλιστα ορισμένα 3,5 χρόνια έχουν ελέγχου στα σύνορα. Αυτό είναι ε, παράνομο και δυσανάλογο. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι για κάτι τέτοιο. Το Σέγγεν είναι υπό απειλή. Το να εγκαταλείψουμε το Σέγγεν θα προκαλέσει απώλεια 18 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για την Ένωση. Ε, δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Καμία χώρα δεν μπορεί να πληρώσει αυτό το λογαριασμό. Έχουμε κανόνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς οποίους μπορούμε να αποκαταστήσουμε την χαμένη εμπιστοσύνη ε, των πολιτών στην Ένωση και να έχουμε κυκλοφορία χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Παρά τα προβλήματα στις ε, διαπραγματεύσεις, ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βοήθησαν αρκετά για να φτάσουμε σε συμβιβασμό. Τα κράτη-μέλη μπλοκάρισαν οποιαδήποτε πρόοδο μάλιστα για συμφωνία ως εισηγήτρια, ως ε, πολίτης, ως Σλοβένα και ως Ευρωπαία καταδικάζω το Συμβούλιο και τη στάση του. Είναι απαράδεκτο ε, λόγω των εσωτερικών πολιτικών ε, συσχετισμών ε, να, παίρνουμε, να κρατάμε όμοιρο το Σέγγεν. Το status quo είναι βολικό για την Κομισιόν στο βαθμό που υπάρχει επιτάπητος η νομοθετική πρόταση και δεν παίρνει δράση, δεν ε, προσφέρει στο δικαστήριο εναντίον αυτών των κρατών μελών. Ε, θα ήθελα να δείξουμε εμείς με την ψηφοφορία μας σήμερα στους πολίτες ότι ενδιαφερόμαστε για την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαγιόν. Ψηφίζουμε. Ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στο, στην πρόταση ψηφίσματος σε τη ε, βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε μια πρόταση ψηφίσματος, ψηφίπε κατά, αποχές εγκρίνεται. Α, αυτό χειροκρότημα ήτανε. Καλά. So, wir kommen jetzt zur letzten Abstimmung. Ε, τελική ψηφοφορία, τελευταία μάλλον. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο. Η κατάσταση ήταν τεταμένη και πολύ σπαραξικάρδια και θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά για την κατανόησή τους τους συναδέλφους οι οποίοι τήθηκαν στις προηγούμενες αμπλόκ ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας που επιλέξαμε αυτή την ε, οδό. Λοιπόν, έκθεση Νετφέλτ, ονομαστικά αρχίζει τώρα η ε, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους σας. Και όπως πάντα θα σας παρακαλούσα να αποχωρήσετε συντόμως για να μπορέσουμε να περάσουμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Ansonsten werde ich nach einiger Zeit die Kollegen. μετά από λίγο θα αρχίσω να λέω ονόματα συναδέλφους που γνωρίζω προσωπικά και είναι ακόμα στους διαδρόμους. Dann darf ich. Λοιπόν, αρχίζω να λέω ονόματα. Μποστινάρου, παρακαλώ. Τον συνάδελφο Μαρινέσκου, Πέρο, Ζαμπάνσκι. Wen kenne ich denn noch? Ποιον άλλον ξέρω. Α, De Jong. Der Herr Kollege Jip. Jip. Herr Kollege Zwiefka. Zwiefka. Frau Kollegin Grostetz, Frau Kollegin Niebler. Die wollen alle ins Protokoll. Καλά, όλοι θέλουν να δουν τα ονόματά τους στα πρακτικά. Γκροστέτ, Νίμπλερ, Ινετφέλτ. Herr Kollege Sarius Wolski. Ach, dem Herrn Kollegen Zambatski habe ich Unrecht getan, der hat ja das Wort. Τον οδήγησα τον κύριο Τζαμπάσκι γιατί ε, καλά κάνει και κάθεται και είναι και όρθιος εδώ γιατί θα πρέπει να πάρει το λόγο για επεξήγηση ψήφου. Κύριε Ρανζέλ. So, jetzt kommen wir zu den Stimmen. Λοιπόν, τώρα περάμε σε εξηγήσεις ψήφου. Έκθεση Κίλωνεν. Για τις οδικές μεταφορές, ο κύριος Σαμπάσκι έχει ε, πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ, συναδελφοί. Ε, εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή αυτή η έκθεση δεν απεικονίζει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών από τις μικρές χώρες στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό την καταψήφισα ήταν επονίδιστη η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Τσαμπάσκι. Κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ συνάδελφοι τελικά αποφάσισα να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση προσπαθώντας να βρω έτσι μια ισορροπία. Ήταν δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμό. Ε, εύχομαι όλοι οι οδηγοί να έχουν καλέ συνθήκε οδήγηση, ε, ωραίο περιβάλλον εργασία και αξιόπιστε μεταφορέ. Οι οδικέ μεταφορέ είναι πυλώνα τη εσωτερική αγορά. Χωρί αυτέ, η ελεύθερη κυκλοφορία δεν θα ήταν αυτή που ξέρουμε σήμερα. Η ανεπαρκής εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων θα μπορούσε να υποσκάψει τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτό το νόμισμα, ε, δύο όψεις του νομίσματος, αλλά τελικά είμαι υπέρ του συμβιβασμού που βγάζει ε, αυτό το τμήμα της εσωτερικής αγοράς ε, από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτιώσει στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Σόιδροβα. Παρακαλώ συνάδελφοι. Σάρβαμα. Ποιον άλλον βλέπω γνωστό. So, jetzt spricht Herr Kollege Mamikin. Ο κύριος Μαμίκινς τώρα. Uh, thank you very much, dear... Ευχαριστώ συνάδελφοι σε ό,τι αφορά τον, τις μεταφορές και τον τουρισμό. Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι η νομοθεσία που υιοθετούμε είναι υπέρ των χωρών και της χώρας μας της Λετωνίας. Αυτή η σημαντική οδηγία για την απόσπαση των οδηγών θα ήταν τμήμα ενός πακέτου που σέβεται και τα τις πτυχές αγοράς αλλά και τις κοινωνικές πτυχές. Λυπάμαι που είναι περισσότερο υπέρ της αγοράς και λιγότερο υπέρ των κοινωνικών θεμάτων στις οδικές μεταφορές. Φυσικά δεν πρέπει να προωθήσουμε τι παράνομε πρακτικέ και πρέπει να μειώσουμε το διοικητικό άχθο, αλλά οποιαδήποτε νομοθεσία περνάμε εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη. Αλλά η ιδέα τη ε, ίση αμοιβή για, ίση, για τι ίδιε ε, υπηρεσίε σε ό,τι αφορά το καμποτάζ είναι θέμα κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ίδιοι κανόνε ε, ισχύουν για το πώς πληρώνεται ε, ένας οδηγό ο οποίος παραδίδει αγαθά σε μια ξένη χώρα όπως και ο οδηγό που παραδίδει αγαθά στη δική του χώρα. Άρα καταψήφισα λοιπόν αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Μπορεί να είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον για το γεγονός ότι αφορά ε, ένα κείμενο για την αγορά, όπου επιβάλλονται περισσότεροι κανόνες ε, στον ιδιωτικό τομέα, μειώνεται η ανταγωνιστικότητα και από την ε, διείσδυση ε, ξένων δυνάμεων. Είναι κακό ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν μικρά περιθώρια κέρδους. Μια και είναι η δική μου ομιλία, θα ήθελα να υποφεληθώ για να σας ευχαριστήσω εσάς κύριε Βίλαν, που πάντα ήσασταν αμερόληπτος, σοφός και αποτελεσματικός α, αντιπρόεδρος. Ε, σας αξίζει αυτός ο θόκος που κάθεστε και αν αυτή είναι η τελική μας συνομιλία θα ήθελα να αποχωριστούμε σαν φίλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαράν. Κανονικά δεν σχολιάζω τέτοια θέματα. Αλλά σπάνια μπορεί, μπορεί σπάνια να συμφωνούσαμε, αλλά πάντα εκτιμούσα την κοινοβουλευτική σας δουλειά. Και ποιος ξέρει, μπορεί να μην ήταν και η τελευταία σας ομιλία. Δεν βλέπω ότι η συνάδελφο Γιασλοβιέτσκα. Οπότε ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Κίλονεν και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Βάντεν Κάμπ ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγηση, κατώτατα όρια για τα διαλύματα, περίοδοι ανάπαυση και εντοπισμό μέσω ταχογράφων. Και πάλι ο κύριο Ζαμπάσχη, έχει το λόγο. Πρόεδρε, συνάδελφοι, αυτή η έκθεση, όπω και η προηγούμενη έκθεση, είναι άδικε για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες της περιφέρειας. Η, η πρόταση θέλει το εξής όλες οι εταιρείε από τις περιφερειακές χώρες να πτωχεύσουν και να φύγει ε, και να μετεγκατασταθούν όλες οι εταιρείε εν στη Δυτική Ευρώπη. Ε, αυτό είναι κατά της ελεύθερης αγοράς, κατά του ελεύθερου ανταγωνισμού, είναι προστατευτισμός 100% ε, από πλευράς Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Με αυτή την έκθεση Είμαστε κατά τη ιδέα Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλες οι χώρες έχουν σημασία και τα συμφέροντά τους έχουν σημασία. Γι' αυτό την καταψήφισα. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθηκε η ψηφοφορία ήταν απαράδεκτος. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσχη. Η κυρία Σόντροβα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας εξηγήσω γιατί τελικά υπερψήφισα αυτή την έκθεση δεν αφορά μόνο τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση, αλλά την ασφάλεια στους δρόμους μας. Αποφάσισα να υποστηρίξω την πρόταση και θα ήθελα οι οδηγοί να έχουν το δικαίωμα να περνάνε το Σαββατοκύριακό τους με τις οικογένειές τους και να έχουν και έναν ελάχιστο χρόνο ανάπαυση. Επίσης είναι λογικό να έχουμε ε, και χώρους ε, παρκαρίσματος με τον απαραίτητο εξοπλισμό, γιατί αυτές οι συνθήκες δεν μπορεί να τις εξασφαλίσει απλώς ο εργοδότης. Ε, πρέπει να υπάρχει πανευρωπαϊκή υποδομή για κάτι τέτοιο. Και σήμερα είναι τραγική η κατάσταση. Θα πρέπει να φτιάξουμε περισσότερους χώρους για παρκάρισμα, θα πρέπει να έχουμε έξυπνους ταχογράφους και όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε χάρη στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σόντροβα. Ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, συμφωνώ ότι οι συνθήκες εργασίας των οδηγών πρέπει να βελτιωθούν. Με τους νέους κανόνες αν δημιουργήσουμε, θα πρέπει να είναι υποφελή ε, για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για την Δυτική Ευρώπη. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Οι οδηγοί από την Ανατολική Ευρώπη θα δυσκολευτούν να κρατήσουν τη δουλειά του. Είμαι κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ και λυπάμαι που η έκθεση είναι σχεδιασμένη για να τιμωρήσει πολλού ανθρώπου από αυτέ τι χώρε. Μιλάμε για το πεπρωμένο των τριών εκατομμυρίων εργαζομένων που διακυβεύεται. Θέλω ε, να υπάρχει ελευθερία στην, ε, στο στην κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και της παροχής ε, υπηρεσιών χωρίς να υποσκάπτουμε τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Δεν θέλω να αφήσουμε χωρίς προστασία, ούτε να πετάξουμε έξω από την ενιαία αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους εργαζομένους από την Ανατολική Ευρώπη. Γι' αυτό καταψήφισα. Ο κ. Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Δεν ψήφισα υπέρ της ε, έκθεσης αυτής, ούτε κατά, απήχα. Γιατί αυτή η έκθεση ενισχύει τα παλιά σύνορα του σιδηρού παραπετάσματο μεταξύ των παλιών και των νέων κρατών μελών της Ένωσης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι ασφάλειες οδικές μεταφορές. Προφανώς. Γιατί οι οδικές μεταφορές αυξάνονται, οι συνθήκες στους δρόμους γίνονται όλο και χειρότερες και οι καλές συνθήκε εργασίας για τους οδηγού είναι πολύ σημαντικέ. Νομίζω ότι αυτό που είναι αποδεκτό είναι η εργαζόμενοι αυτοί να έχουν χρόνο ανάπαυση στι καμπίνε του, να περνάνε χρόνο με τι οικογένειέ του. Σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό που είναι απαράδεκτο είναι το πώ ψηφίσαμε και το πώ συζητήσαμε του εμβιβασμού. Γι' αυτό δεν υποστήριξα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόλτσακ. Τελειώσαμε την έκθεση Φαδενκάμπ και τώρα προχωρούμε σε επεξηγή ψήφου τη έκθεση Ερτούκ με θέμα την προσαρμογή τη εξελίξη στον κλάδο οδικών μεταφορών. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για μια ακόμη φορά Οπότε και πέρα του τη συζήτηση και επεξήγηση ψηφία το πακέτο αυτό, πρέπει να σα πω ότι καταψήφισα την έκθεση Ερτούκα στο πλαίσιο τη δέσμη μέτρων. Θεωρώ ότι πρόκειται κατάφορη παραβίαση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού. Όταν θέλουν στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, δυτικέ εταιρείε να πουλήσουν, υπάρχουν τεράστια σούπερ μάρκετ και έρχονται και πόλουν τα προϊόντα του. Όταν όμω Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία θέλουν να εργαστούν ε, στη Δυτική Ευρώπη, οι πόρτε είναι κλειστέ. Αυτό είναι άδικο. Και αντιβαίνει στην ίδια την αρχή της ενιαία και ελεύθερης αγοράς ε, που πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή ψηφοφορία διεξήχθη με ε, αναξιοπρεπή τρόπο και παραβιάστηκαν πολλοί κανόνες. Όμως ήταν η πιο σκανδαλώδη ψηφοφορία που έλαβε ποτέ χώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν διχασμένοι 50-50 οι βουλευτές, δεν υπήρχε πλειοψηφία, τελικά επικράτησαν οι λομπίστες γιατί αυτοί επηρέασαν και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν αυτή την εξέλιξη Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Συναφέ Τζαμπάσκι. Κυρία Σόντρεβα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ε, του πακέτου αυτού είχε βρεθεί συμβιβασμό ε, στο πλαίσιο της Επιτροπής Μεταφορών και ήταν ε, η μόνη από τις τρεις εκθέσεις ε, όπου αυτό έγινε, από, έγινε δυνατόν. Έτσι θα είναι λίγο πιο εύκολο ο ερχόμενο τριμερής διάλογος. Το καμποτάζ ήταν πάντο κάπως διαφορετικό από τις διεθνείς οδικέ μεταφορέ ή τα διάφορα πρότυπα. Υπάρχει εδώ άμεσο ανταγωνισμό με τους μεταφορείς στις εγχώριες αγορές. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι κανόνες ε, να είναι τέτοιοι ώστε να μην διαταράσετε το σύστημα των οδικών μεταφορών ούτε ε, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που εξαρτάται ακριβώς από την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν όλο το πακέτο να αξιολογηθεί όμως Εκτιμώ ότι δεν τίθενται μόνο για το καμποτάζ όρια στην έκθεση, αλλά περιλαμβάνονται και μέτρα κατά των ε, εικονικών εταιριών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι προληπτικό μέτρο που θα μας επιτρέψει από αυτήν καταχρήση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευχαριστούμε, κυρία Σόντροφα. Ο κύριος Μάθιος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την πρόταση αυτή, διότι όπως και πολύ συχνά εδώ σε αυτό το μέρος, ουσιαστικά επιβαρύνει υπερβολικά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δύσκολα μπορούν να το αντέξουν το βάρος αυτό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι όμιλοι μπορούν να πληρώνουν τους λομπίστες που περιμένουν έξω από την πόρτα και επηρεάζουν το νομοθετικό έργο. Δυστυχώς αυτό φοβάμαι ότι είναι ένα ακόμη παράδειγμα Βλέπουμε ότι τελικά ε, η νομοθεσία είναι κομμένη και αραμένη για τις μεγάλες επιχειρήσεις που ε, επομιστούν αυτό το έξτρα κόστος. Δεν μπορούν να το κάνουν όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό τις θέτουμε σε ε, μειονεκτική θέση και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δυσανάλογα μπορούν να επηρεάσουν τέτοιοι κανόνες επιχειρήσεις εξού και ψήφισα κατά του μέτρου για να στηρίξω τις μικρές εταιρείες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μάθιο. Επόμενο ο συνάδελφο κύριο Πόλτσακ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση διότι τελικά καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν πραγματικό συμβιβασμό. Και αυτό διαφοροποιεί αυτήν την έκθεση από τις δύο προηγούμενες μέτρων για την κινητικότητα. Οι οδικές μεταφορές ε, αναπτύσσονται, υπάρχουν νέες τεχνολογίες, αυτόνομη οδήγηση και τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών. Η Ευρώπη όμως ε, υπολείπεται άλλων χωρών και θα πρέπει να εξελιχθούμε κι εμείς. Πάντω η έκθεση ευθυγραμμίζεται με τις δικές μου επιθυμίες, εξού και την υποστήριξα. Σε ό,τι αφορά τώρα το καμποτάζ, νομίζω ότι θα πρέπει να καλυφθεί με νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πόλτσακ. Ολοκληρώνονται εδώ η εκθέση του. Κυρία Γιασλοβέτσια, ε, ε, ε, πρόκειται να μιλήσετε προηγουμένως. Μπορώ να σας δώσω το λόγο στο τέλος, αλλά όχι τώρα. Προχωρούμε στην επόμενη έκθεση. Μπούζεκ. Κοινή κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Κυρία Γιασλοβιέσκα, δεν θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριος Μαμίκινς έχει το λόγο. Thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν μπόρεσα να συμφωνήσω με τον τρόπο με τον οποίο ε, επινοήθηκε αυτή η οδηγία. Καλά, να διακόψω. Κύριε Γιασλοβιέσκα, σας ανακαλώ στην τάξη. Κύριε Μαμίκινς, έχετε το λόγο. Thank you. Thank you, President. Once again. I could... Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ με τη σύλληψη της ίδια αυτή της οδηγίας. Κατά την άποψή μου, οποιοδήποτε κανόν ε, ε, για, για την ε, ενέργεια θα πρέπει να είναι σαφής και να μην στρέφονται κατά ενό ή άλλου έργου και κατανοείται ότι γίνεται λόγος για τον αγωγό φυσικό αερίου Nord Stream 2 από τη Ρωσία προς τη Γερμανία. Ε, ε, αυτή η αγωγή από ή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα της ενεργειακής ασφάλειας και της υποδομής μας και επιτρέπει σε τρίτες χώρες και άλλους προμηθευτές και εταίρους μας να είναι τμήμα ε, της αρχιτεκτονικής μας αυτής της ενεργειακής και φοβούμε ότι η οδηγία αυτή έχει κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι για τον ανταγωνισμό ε, θα πρέπει ε, οι ε, παράγοντες που έχουν δεσπόζουσα θέση και οι μικροί φορείς να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να μην την πληρώνουν τελικά οι καταναλωτές και να μην πέφτουμε θύματα σε, της αντιρωσικής ρητορικής. Εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Μαμίκινς. Κυρία Γιασλοβιέσκα, αν δεν σταματήσετε αμέσως θα σας απομακρύνω από το εμικύκλιο. Το λόγο έχει τώρα ο ε, συνάδελφος Στρογεύσκη. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ίσως η κυρία Γιασλοβιέτσκα ε, έχει να δώσει κάποια εξήγηση για το λόγο της απουσίας της προηγουμένως. Δεν ξέρω. Δεν θέλω εγώ να παρέμβω σε αυτό μήπως να της δίνατε το λόγο, να της επιτρέπατε να μας εξηγήσει. Ε, ωραία. Κυρίες και κύριοι, ε, γίνεται λόγος εδώ για την ασφάλεια. Ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και κατανοώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχουν οι εταιρείε ασφάλεια δικαίου. Και χαίρομαι που καταλήξαμε σε 15 θετικούς συμβιβασμούς και βρήκαμε λύσεις. για τα νέα δίκτυα εντός, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ γίνεται λόγος για τους ε, αγωγούς φυσικού αερίου και για την αποσύνδεση του καθεστώτος ιδιοκτησίας από τη μεταφορά. Ε, τέλος, ε, το πεδίο εφαρμογής τη οδηγία. Όλα αυτά είναι σωστά ε, και κάποιες εξαιρεσει που εισήχθησαν δεν θα κάνουν τίποτα άλλο παρά να βοηθήσουν το σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Στρογγεύσκη και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και εγώ υποστήριξα την έκθεση αυτή. Όπως και προλαλής σας κατανοώ και εγώ ότι όταν δημιουργούμε μια ενεργειακή ένωση, ένα τμήμα του κλάδου ε, θέλει να εξασφαλίσει και ε, ανεξαρτησία από τους προμηθευτές. Είναι και κάποια γεωπολιτικά ζητήματα. Η Ρωσία μπορεί να είναι απειλή ε, για μας και μεγάλη μας εξάρτηση, μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ενέκρινα την πρόταση αυτή που επεκτείνει τους κανόνες και τις υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου και αφορά και το επίμαχο ε, έργο Nord Stream 2. Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν και για τις ρωσικές εταιρείες, ε, την Gazprom ουσιαστικά που δεν θα μπορεί να καταχράτε ε, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που έχει την αγορά. Και έτσι θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα διαπούν τις δραστηριότητες και της Gazprom. Ευχαριστώ κύριε Πόσπιση ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ενεργειακή Ένωση είναι κρίσιμο στοιχείο του μέλλοντός μας. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε την γεωπολιτική, την ασφάλεια, Έχουμε χρέος να το κάνουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ε, διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού, όχι μονομέρεια. Γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε με κοινούς στόχους, ειδικά τους γεωπολιτικούς. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω αυτή την πρόταση να διαχωρίσουμε την ιδιοκτησία από τη διανομή. Ελπίζω να δουλέψει αυτό στο μέλλον Η λειτουργία του κλάδου του φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι τμήμα αυτή τη Ενεργειακή Ένωση και γι' αυτό η πρόταση είναι πολύ θετική. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής και συγχαίρω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε, τον πρώην πρόεδρο Μπούζεκ και την Κομισιόν γιατί συνεργάστηκαν για να πετύχουν ένα καλό αποτέλεσμα για όλους μας. Είναι καλή ιδέα όλοι οι αγωγοί να διέπονται από τους ίδιους κανόνες, οι αγωγοί που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά και το North Stream αυτό και άλλους αγωγούς. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το 77% της, ε, του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην ε, Ένωση περνάει μέσα από αυτούς τους αγωγούς. Στο μέλλον, όλοι οι κανόνες εφαρμόζονται ίδια ε, σε αυτούς που είναι στην Ένωση και σε αυτούς που μπαίνουν στην Ένωση. Κάναμε μια προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε την ενεργειακή αγορά, να ολοκληρώσουμε την Ενεργειακή Ένωση και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για τη δουλειά που κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Κέλλη. Προχωρούμε, αφού τελειώσαμε την έκθεση Μπούζεκ, στην έκθεση ΜΑΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ο κύριος Σόσνιρτς. Εγώ καταψήφισα αυτή την έκθεση. Κοιτάξτε το σημείο 422α και θα δείτε ότι ακόμα μια φορά Είμαστε στο χώρο του παραλόγου. Με αυτό το άρθρο ζητάμε ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Τι λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό. Καταλαβαίνω και τις κυρίες, τις ευρωβουλευτίνες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υπερψήφισαν την έκθεση αυτή. Τις φαντάζομαι να μπαίνουν τώρα σε αλληλευτικά σκάφη. Μια τέτοια μακροσκελής και ανιαρή έκθεση θα έπρεπε να καταψηφιστεί και εγώ την καταψήφισα τουλάχιστον. Ευχαριστώ κύριε Σόσνες. Ο κύριος Κέλλη τώρα. Ευχαριστώ. Το σύστημα ε, που ισχύει σήμερα ήταν πολύ περίπλοκο. Ε, δεν δίνει παρά τη χρηματοδότηση αυτούς που το ε, χρειάζονται. Ε, χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο ευέλικτη πρόσβαση ε, στην αποζημίωση του ταμείου σε περίπτωση που σταματήσει οριστικά η αλληλευτική δραστηριότητα. Και οι νέες διατάξεις θα πλουστεύσουν το σύστημα ε, και θα υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στα κονδύλια. θα υποφεληθούν πολύ οι Ιρλανδοί αλληλείς, καθώς και τα νησιά μας, εξού και οι τροπολογίες. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ε, υπάρχουν κάποια προσχεδιασμένα μέτρα για τους κανόνες επιλεξιμότητας. Επίσης, ε, υποστηρίζονται οι επενδύσεις και βελτιώνεται η ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας το, του πληρώματος στο κατάστρωμα και στα σκάφη. Αυτά, γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε την έκθεση ΜΑΤΟ. Ακολουθεί τώρα η έκθεση ΝΤΕΠΡΕΦ ενίσχυση τη ασφάλεια των δελτίων ταυτότητα και των εγγράφων διαμονή που εκδίδονται για του πολίτε τη Ένωση. Ο κ. Δρουγεύσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 100 περίπου διαφορετικών ειδών δελτία ταυτότητας και 200 διαφορετικά έγγραφα ε, είναι πολλαπλάσιο ο αριθμό αυτό των κρατών μελών. Γι' αυτό ε, χαίρομαι για τη συμφωνία που επετεύχθη στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, για να υπάρξει μια εναρμόνιση των ταξιδιωτικών εγγράφων και των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονή. Ε, για την συλλογή βιομετρικών ε, στοιχείων και δεδομένων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η γνησιότητα των εγγράφων αυτών. Υπερψήφισα την έκθεση γιατί μου άρεσε αυτό το στοιχείο της εναρμόνισης. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, έχουμε πενταετή διάρκεια των ταυτοτήτων και τα λοιπά, ανάλογα με την ηλικία των πολιτών είναι σημαντικά τα έγγραφα αυτά κατά την άποψή μου, ιδιαίτερα για κάποια κράτη-μέλη. Ε, γιατί ορισμένα χάνονται κιόλας ή καταργούνται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ υποστήριξα τη συγκεκριμένη έκθεση παρότι υπήρξε έντονη συζήτηση στη χώρα μου όμως θεωρώ παρόλα αυτά ότι μπορεί αυτή η έκθεση να βοηθήσει στο να είναι πιο δύσκολη η πλαστογράφηση των δελτίων ταυτότητας. Τα ελάχιστα δε πρότυπα ασφαλείας είναι θετικά και τα περί βιομετρικών απαιτήσεων που ενισχύονται. Αυτά θα βελτιώσουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στην Ένωση. Θα βελτιώσουν όμως ταυτόχρονα και την ασφάλεια και θα μειώσουν τις περιπτώσεις ανθρώπων που κυκλοφορούν πλαστά διαβατήρια. Δεκάδες εκατομμύρια πολιτών θα έχουν πλέον πιο ασφαλείς ταυτότητες και αυτό είναι πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνει ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα τον κανονισμό που πιστεύω ότι θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων και την εφαρμογή ελάχιστων προτύπων για άδειε διαμονή που εκδίδουν τα κράτη-μέλη ή για τις ε, ταυτότητες των ε, πολιτών. Πάνω από 20 ε, εκατομμύρια εργάζονται και ζουν αλλού και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία περνούν τα εξωτερικά σύνορα, δισεκατομμύρια και αυτά τα πλαστά ε, διαβατήρια ταξιδιτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτε, εγκληματίε. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών μέσω πιο ασφαλών ε, ταυτοτήτων και καρτών παραμονή που εκδίδονται για τα άτομα αυτά και τα μέλη των οικογενειών. Του χαιρετίζω τι προσπάθειε καταπολέμηση τη απάτη λόγω πλαστών εγγράφων ε, και πλαστοπροσωπία είναι ένα τομέα αυτό που θα ήθελα η Ένωση να κάνει περαιτέρω δουλειά, ώστε να μην ε, υποφέρουν αθώοι από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε και λέει ο πρόεδρο. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτή και περνάμε στην έκθεση κυρία Αγιού για τη διαχείριση της ασφάλεια των οδικών υποδομών. Μάθιους είναι ο πρώτο ομιλητή. Αύριο είναι μέρα που πάμε στη δουλειά μας με τα πόδια. Το έκανα σήμερα, θα το κάνω και αύριο. Το βάδισμα είναι πάρα πολύ ευχάριστη δραστηριότητα, σωματική άσκηση, ε, βάζει, φέρνει το γιατρό μακριά, ε, βοηθάει στην ευεξία. Με τις οδικές υποδομές που έχουμε όμως ε, παραγνωρίζονται οι ανάγκες των πεζών, γι' αυτό με πολύ χαρά υπερψήφισα την έκθεση αυτή, όχι μόνο διότι λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πεζών, όμως όμως ε, ταυτόχρονα αναγνωρίζει πως πρόκειται για έναν τομέα όπου τα μεμονωμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την πρωτοκαθεδρία και να μην υπάρχει εναρμόνιστον των πάντων γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη με τοπικές συνθήκες, τοπικές προτιμήσεις. Άρα και για τους δύο αυτούς λόγους θα στηρίξω την έκθεση και περιμένω με υπομονησία το πώς θα ψηφίσουμε για τους αυτοκινητοδρόμους για να είναι και αυτοί πιο φιλικοί Ευχαριστώ, ο κύριος Μάιερ. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την έκθεση αυτή για τη βελτίωση της οδικής ασφάλισης, ασφάλειας των οδικών υποδομών. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα ε, για το ε, πρόβλημα που έχουν τα φορτηγά που τρακάνουν σε χαμηλές γέφυρες και στην εκλογική μου περιφέρεια. 120 ε, φορές έχουν χτυπήσει μια γέφυρα που έχει ύψος τριών μέτρων τα τελευταία δύο χρόνια και συνεχίζει ακόμη παρόλο που έχουν βγάλει μια τεράστια και πολύ ωραία προειδοποιητική πινακίδα και είναι πολύ ακριβώς ο λογαριασμός για τους οδηγούς φορτηγών και τους επιβάτες. Υπάρχουν υψηλή τεχνολογία και χαμηλή τεχνολογία ε, που μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή ε, να κρέμεται κάτι πριν από τη γέφυρα που να χτυπάει στην οροφή του φορτηγού και να προειδοποιεί. Ευχαριστώ κυρία Μάια. Τελειώσαμε με την έκθεση του. Και τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Σίντφελτ, θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος. Ο κύριος Μπενίτο Σιλουάγα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταψηφίσαμε το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν. Εσείς και η Θιουδαδάνο και το ΕΛΚ ε, ψήφισαν ναι. Ναι στι συντάξει των πλουσίων. Γιατί αυτές ε, θα είναι οι συντάξεις. Ε, και εσείς έχετε όλο και πιο πλούσιες ε, ε, συντάξεις. Στο μεταξύ ε, μειώνονται οι δημόσιες συμβάσεις που στηρίζουν τους πιο φτωχούς και την οικονομία και πολλές οικογένειες. Μιλάτε για τις ιδιωτικές συντάξεις, τις οποίες πληρώνουν με τις συνεισφορές τους διάφοροι για να στηρίζουν τους πλούσιους. Όσοι δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν ιδιωτική σύνταξη, α κάνουν τι νομίζουν. Ε, οι περικοπέ τη ε, λιτότητα δεν ε, οδηγεί στην φτώχεια και στην. Στην πραγματικότητα όμως τις χρησιμοποίησατε την κρίση εσείς για να επιβάλλετε το νεοφιλελεύθερο μοντέλο σας. Οι δίκες συντάξεις δεν πουλούνται. Θα πρέπει να τις υπερασπιστούμε. Ευχαριστώ κύριε Στρογεύσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ διαφωνώ με τον Λίσαντα. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση αυτή και οι συμβιβασμοί είναι πολύ θετικοί. Ειδικά δύο από αυτούς τους συμβιβασμούς. Πρώτον, οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν ένα συνταξιδοτικό προϊόν διασυνοριακά. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Εν συνεχεία, η μείωση του κόστους από το 1,5% στο 1% θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό. Όλη η έκθεση λοιπόν κατά την άποψή μου είναι θετική και θέλω ε, τρία χρόνια μετά την υιοθέτηση ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Στρογεύσκη. Τελευταίος τώρα ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υποστήριξα αυτή την έκθεση γιατί είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τις ενδιάμεσες γενιές ούτω ώστε να βελτιώσουν την κατάστασή τους όταν φτάσουν ε, σε, στο γύρας. Οι νεαροί, οι Ευρωπαίοι, πολύ σπάνια αγοράζουν ε, ιδιωτικές συντάξεις, αρχίζουν να ε, συνεισφέρουν ας πούμε, σε επικουρικά ταμεία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δημιουργήσει νέα ελκυστικά προϊόντα για το, την περίοδο του γύρατος. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες φιλοδοξίες. Θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες φοροαπαλλαγές, Φερρυπίν. Ο συνάδελφο εξεβονίμων είπε ότι αυτό υπάρχει ήδη, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό ακόμα. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικά αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόσπισελ. Ολοκληρώνονται εδώ επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Netfeld. Έχουμε τώρα ακόμα μια επεξήγηση από προηγουμένω από την έκθεση Κίλονεν και θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Εσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα σέβομαι, Πρόεδρε, πρέπει να το πω αυτό και εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε στο Κοινοβούλιο. Ήθελα να πάρω το λόγο γιατί ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία μου όταν συζητήθηκε η έκθεση αυτή η Κιλόνεν. Τα τελευταία 7 χρόνια εγώ ασχολήθηκα με την απόσπαση των εργαζομένων. Ζητώ Ξανά συγγνώμη και μπορώ να πω, φαντάζομαι τώρα, αυτά που ήθελα να πω εξ αρχής. Το πακέτο κινητικότητας που υιοθετήσαμε δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί επαρκώς. Υπάρχει δημαγωγία, υπάρχει προστατευτισμός, υπάρχουν πολλά συναισθήματα που χρησιμοποιήθηκαν, ας πούμε, ε, για να διαμορφωθούν ε, τα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα για τους οδηγούς, ε, για τις και τα επιχειρήματα των εταιριών έχουν αγνοηθεί. Γι' αυτό λοιπόν το πακέτο αυτό και το, τα κείμενα αυτά είναι ό,τι χειρότερο έχει υιοθετήσει ποτέ το Κοινοβούλιο. Το έγγραφο αυτό θα καταστρέψει τις διεθνείς μεταφορές στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν τη λυπητερή. Αισθάνομαι ντροπή που συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία και καταψήφισα το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιασλοβιέτσκα. Ολοκληρώνω την επεξηγήση ψήφου εδώ. Τα συνοπτικά πρακτικά τη παρού συνεδρίαση θα υποβληθούν προ έγκριση στο Κοινοβούλιο στην επόμενη και αν δεν διαφωνείτε, τα κείμενα που εγκρίθηκαν και τι προτάσει ψηφίσματο θα τα διαβιβάσω αρμοδίω στα αρμόδια πρόσωπα και όργανα. Στο τέλο αυτή τη μήνυ συνόδου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλε τι υπηρεσίε και σα εύχομαι καλή επάνωδο, καλή σα όρεξη και ευλογημένη ε, διακόπτεται ε, ε, η σύνοδος, η κοινοβουλευτική περίοδος μάλλον και λίγη συνεδρίαση.